κύριο Έτσιο Περίλο, ο οποίο θα λάβει το λόγο εκ μέρου τη νομική υπηρεσία. Γι' αυτό θα περιμένουμε λίγο λεπτά ακόμα πριν ξεκινήσουμε. We're getting started. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Καταρχάς, να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Δεν έγινε καμία πρόταση αλλαγής για την ημερήσια διάταξη. Επομένως, αν κάποιος δεν έχει αντίρρηση για την ημερήσια διάταξη, εγκρίνεται και περνάμε στο πρώτο Έχουμε λοιπόν το θέμα που σχετίζεται με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Προστασίας. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Έχουμε μια κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών ε, ΛΥΜΠΕ ε, Πολιτικών Ελευθεριών και της Επιτροπής Γυναικών. για την πρωτοβουλία αυτή που προήλθε από πλευρά Συμβουλίου. Πιο συγκεκριμένα, δύο κράτη-μέλη υιοθέτησαν μια πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. ως εφαλτήριο χρησιμοποιούμε το γεγονός ότι η προστασία των θυμάτων είναι προτεραιότητα στην ε, ε, ποινική πολιτική των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για αυτή την πρωτοβουλία θα πρέπει να έχουμε κατάλληλους μηχανισμούς προκειμένου να προστατεύσουμε τα θύματα της βίας, βίας ε, κατά του φίλου ή οποιασδήποτε απόπειρας ε, εγκληματικής ε, που παραβιάζει την φυσική ελευθερία, την ζωή κάποιου από οποιαδήποτε χώρα ή οποιοδήποτε κράτος μέλος και αν προέρχονται. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης ε, και ασφάλειας. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης και το ίδιο διαπιστώσαμε και στον ορισμό του προγράμματος δράσης, ε, το οποίο θα ε, χρησιμοποιήσουμε για την εξέλιξη του προγράμματος της Στοκχόλμης. Γι' αυτό ακριβώς αυτή η πρόταση οδηγίας προσπαθεί να καθορίσει τρόπους προστασίας ένα μέσο προστασίας το οποίο θα μπορεί να εφαρμόζεται και στο κράτος μέλος στο οποίο εκδίδεται η εντολή προστασίας αλλά και σε οποιοδήποτε άλλος κράτος μέλος το θύμα ενδεχομένως να αποφασίσει να μετικήσει. Ο πολιτικός στόχος της πρωτοβουλίας ε, την χάνει ευρύτατη συνένεση μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και ακριβώς Συζητείτε και έχουν προκύψει και κάποιες ε, νομικές ε, και ε, πολιτικές ερωτήσεις για τη νομική βάση, για το να δούμε κατά πόσον μπορούμε να καθορίσουμε το θέμα αυτό και προέκυψε μια συζήτηση για τις αμφιβολίες που υπάρχουν για τη νομική βάση για το θέμα αυτό. Ε, και τις εξέφρασε και η Επίτροπος, ε, η Αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Vivian Redding και κατά συνέπεια επειδή είναι πολύ δύσκολο να συμφιλειωθούν ε, αυτά τα διάφορα νομικά συστήματα και υπάρχουν και οι απόψεις του Συμβουλίου Αφενός και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αφετέρου. Γι' αυτό και οι συντονιστές των Επιτροπών ε, ΛΥΜΠΕ και της Επιτροπής Γυναικών αποφάσισαν να ζητήσουν την ε, γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου. Ναι, Ζητήθηκε λοιπόν αυτή η γνωμοδότηση από την νομική υπηρεσία και του ζητήθηκε να μας ε, την παρουσιάσουν πριν από την κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής ε, ε, της κοινή συνεδρίασης μεταξύ των δύο επιτροπών που θα γίνει στις 22 Ιουνίου στην οποία συνεδρίαση θα έχουμε και μια ψήφο προσανατολισμού. Βάσει και του άρθρου 51 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή η συνεδρίαση στην οποία θα συμπροεδρεύουν η κυρία Εύα Μπρίτ, πρόεδρος Επιτροπής Γυναικών και εγώ. Και σε αυτή την κοινή συνεδρίαση θα ακούσουμε την παρουσίαση της νομικής γνωμοδότησης από πλευράς ε, διευθυντή της νομικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του κυρίου Ρέτζιο Περίλο. Θα του δώσουμε τώρα το λόγο προκειμένου να μας παρουσιάσει τη γνωμοδότηση. Αν συμφωνεί και η κυρία Σβένσον, ο συμπρόεδρος, θα ακούσουμε πρώτα τον κύριο Περίλο και στη συνέχεια θα δώσουμε το λόγο στους εισηγητές, στις εισηγήτριες, οι οποίες είναι υπεύθυνε για το θέμα αυτό, η κυρία Ρομέρο Λόπε από πλευρά Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και από πλευρά Επιτροπή Γυναικών η κυρία Χιμένε Μπεθερέλ. Καταρχά, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Έτσιο Περίλο. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους σε όλα τα μέλη των δύο επιτροπών που συνεδριάζουν από κοινού σήμερα περιγράψατε εν συντομία τις πολιτικές προτεραιότητες που συνδέονται με αυτήν τόσο σημαντική οδηγία. Ελπίζω να είμαι και εγώ εξίσου σύντομο για να σας εκθέσω τους όρους που διέπουν τις πολιτικές κατευθύνσεις πολιτικούς προσανατολισμούς που θα μας οδηγήσουν τελικά στην έγκριση αυτής της οδηγίας. Η νομική υπηρεσία εκλήθη να αναλύσει το εξή ερώτημα. Αν το άρθρο 82, παράγραφο 1, εδάφιο Δέλτα της Συνθήκης της Λισαβόνας, συνιστά την ορθή νομική βάση για την έγκριση της οδηγίας για το ΕΠΟ, δηλαδή για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Όπως υπενθυμίζατε ζητήθηκε για τις 28 Ιουνίου αυτή η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας. Ε, στο ενδιάμεσο διάστημα επισπέστηκε η διαδικασία κατά κάποιο τρόπο για διάφορους λόγους. Ε, σήμερα λοιπόν ε, θα σας μιλήσω για την απάντηση που προτίθεται να σας διαβιβάσει η νομική υπηρεσία υπό την επιφύλαξη της γνωμοδότης που θα ακολουθήσει αμελητή. Και για αυτό το λόγο δεν μπόρεσα να δώσω στους διερμηνείς, λέει ο μιλητής, στο κείμενο της παρέμβασής μου και ζητώ συγγνώμη. Θα αναφερθώ σε κάποιες διατάξεις της συνθήκης και θα τις διαβάσω αργά για να διευκολύνω τους διερμηνείς. Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Όπως είπατε πρόεδρε, είναι ένα μέτρο ε, Νέο και ρηξικέλευθο. Στο πλαίσιο του ε, χώρου ελευθερίας, ε, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Ένα τέτοιο νέο και ρηξικέλευθο μέτρο ε, θέτει ευαίσθητα ζητήματα επιτάπητος και διάφοροι όπως και ο υποφαινόμενος ε, φυσικά δεν ισχυρίζονται να έχουν το μονοπόλιο και να κρατούν την απόλυτη αλήθεια. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να βασιστούμε σε αντικειμενικά στοιχεία χωρίς να επισέλθω σε τεχνικού χαρακτήρα λεπτομέρειες για αυτή την οδηγία. Θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας είναι η... ένα μέτρο προστασίας, ε, όπως λέει και το όνομά του. Και προστατεύει κάποιον που εκτίθεται σε κίνδυνο βίας. Επιτρέψτε μου, Πρόεδρε, να γίνω πιο συγκεκριμένος. Δεν χρειάζεται να έχει πέσει θύμα βίας ή ε, ε, βίαιης επίθεσης ε, ή οποιασδήποτε εγκληματικής αξιόπινης πράξης. Φτάνει να έχει εκτεθεί σε ένα κίνδυνο βίας ή επίθεσης σεξουαλικής, ψυχολογικής, ηθικής, οτιδήποτε. Ένα μέτρο προστασίας λοιπόν για κάποιον που εκτίθεται σε κίνδυνο από κάποιον άλλον που έχει θεωρηθεί επικίνδυνος λόγω της συμπεριφοράς του που είναι βίαιη ή επιθετική. Ε, ή που προτίθεται να κάνει μια σεξουαλική επίθεση. Προστατεύουμε κάποιον λοιπόν σε σχέση με κάποιον που ίσως δεν έχει καταδικαστεί αλλά μπορεί να είναι υπόδικος. για να χαρακτηρίσουμε την ε, νομική φύση της Ευρωπαϊκής Εντολής Προστασίας από νομικής πλευράς ε, θα τα δούμε όλα αυτά τα επιμέρους σημεία. Ποιο είναι το άλλο νέο στοιχείο του ΕΠΟ. Είναι ένα μέτρο προστασίας που προστίθεται στα εθνικά μέτρα προστασίας. Ε, το θεμέλιο δηλαδή είναι ένα εθνικό μέτρο προστασίας και από πάνω έχουμε το μόσχευμα το, της Ευρωπαϊκής Εντολής Προστασίας. Εξάλλου εκδίδεται από την ίδια Εθνική Αρχή η Ευρωπαϊκή Εντολή προστασίας ή μπορεί να ζητηθεί από κάποια άλλη ε, αρμόδια εθνική αρχή. Τι γίνεται λοιπόν. Ε, μέσω της Ευρωπαϊκής Εντολής Προστασίας κάποιος, μια γυναίκα ας πούμε, που την χάνει ήδη προστασία σε δυνάμει ενός εθνικού μέτρου στο κράτος μέλος της, αν αποφασίσει αυτή η γυναίκα να μετικήσει σε άλλο κράτος μέλος ε, ή να πάει σε άλλο κράτος μέλος για σύντομη ή για μακρά χρονική περίοδο, μπορεί να ζητήσει από την Εθνική Αρχή που έχει εκδώσει το εθνικό μέτρο να επεκτείνει ε, το μέτρο, όχι να δημιουργήσει κάτι καινούριο, να επεκτείνει την ε, προστασία, την αρχική προστασία στην επικράτεια του κράτους μέλους το οποίο προτίθεται να ταξιδέψει, να μετικήσει, οτιδήποτε. Αυτό είναι το πνεύμα που διέπει την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Επειδή έχει ευρωπαϊκή διάσταση, επιτρέπει να επεκτείνουμε ένα εθνικό μέτρο προστασίας που έχει ήδη αποφασιστεί, έχει ήδη εγκριθεί κατόπιν. Με στην οδηγία θέτουμε και τους ελάχιστους όρους. Είναι ένας νομικός όρος αυτός που χρησιμοποιώ. Και το ΕΠΟ, Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας, ε, ε, εγκρίνεται... σε σχέση με αυτόν που συνιστά τον κίνδυνο. κατά αντιπαράσταση με αυτόν που συνιστά τον ε, κίνδυνο. Ε, και όλα αυτά στο, με στόχο την πρόληψη ε, της διάπραξης μιας αξιόπινης πράξης. Για να περάσω τώρα στη νομική βάση της οδηγίας. Υπάρχουν δύο σχολές, αν θέλετε, οι δύο τάσεις, οι δύο απόψεις για τη νομική βάση. Η μία θεωρεί ότι το άρθρο 82 για την συνεργασία σε ποινικά ε, θέματα δεν είναι η σωστή νομική βάση. Γιατί, διότι η Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας μπορεί να εκδοθεί από εθνικές ε, διοικητικές ε, δικαιοδοτικές αρχές, ε, δηλαδή αρχές που δεν είναι απαραίτητα δικαστικές αρχές. Άρα υπερβαίνει το άρθρο 82 και τη συνεργασία για ποινικά ζητήματα. Οπότε αν θέλουμε να θεσπίσουμε μια οδηγία για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας, ε, είπαν κάποιοι θα πρέπει να πρέπει να περιορίσουμε την οδηγία όταν υπάρχει αδίκημα ε, που θα δικαστεί από έναν δικαστή ποινικού δικαίου και οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο άλλης οδηγίας που θα βασίζεται αυτή τη φορά στο άρθρο 81 που σχετίζεται με την δικαστική συνεργασία σε αστικά θέματα. Αυτή η σχολή λοιπόν θεωρεί ότι ένα μέτρο δεν μπορεί ταυτόχρονα να υπάγεται και στο αστικό και στο ποινικό δίκαιο. Εφόσον αναφέρθηκε σε αυτό και ο Πρόεδρος, ε, σε αυτή τη σχολή. Η σχολή αυτή υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θεωρεί ότι αν θέλουμε ΕΠΟ, Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας, ε, ε, πρέπει να υπάρχει ποινικό αδίκημα. Και αν θέλουμε να προσθέσουμε μέτρα αστικού δικαίου, χρειάζεται άλλη νομική πράξη που θα βασίζεται σε άλλη νομική βάση, δηλαδή το άρθρο 81. Η δεύτερη σχολή αντίθετα θεωρεί ότι το άρθρο 82 εδάφιο δέλτα είναι η σωστή νομική βάση, δηλαδή η διευκόλυνση της ποινική συνεργασίας, γιατί διότι τα ποινικά ζητήματα μέσα στη συνθήκη της ε, Λισαβόνας ε, είναι ε, μια αυτόνομη ιδέα αυθύπαρκτη που δεν συμπίπτει με τα αντίστοιχα ποινικά θέματα σε κάθε κράτος μέλος. Επειδή είναι αυθύπαρκτη λοιπόν αυτή η έννοια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την νομική βάση για να εγκρίνουμε ευρωπαϊκές εντολές προστασίας άσχετα με το αν έχουν εκδοθεί από δικαστικές αρχές ή από αρχές αστικού δικαίου. Βάσει αυτής της δεύτερης σχολής, στην νομική βάση του άρθρου 82 εδάφιο Δ, πρέπει να προσθέσουμε και το εδάφιο Α του 82, για την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων σε ποινικέ υποθέσεις δύο νομικές βάσεις μέσα στο ίδιο άρθρο, έτσι, 82α και 82 δέλτα. Εντάχει αυτά ήταν τα ε, στοιχεία αυτής της ε, ε, νομικής αντιπαράθεσης που μας απασχολεί σήμερα το πρωί. Η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου δεν συμφωνεί με την πρώτη σχολή και ε, συμφωνεί μόνο εν μέρη με τη δεύτερη σχολή σκέψης. Θεωρώ ότι η τωρινή πρόταση οδηγίας για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας εδράζεται όχι μόνο στο άρθρο 82 Δέλτα, είναι η νομική βάση μέσα στο σχέδιο οδηγία και υποστηρίζεται από την νομική υπηρεσία του Συμβουλίου, σε παρένθεση αυτό. Αλλά πρέπει να εδράζεται και στο άρθρο 3 τη συνθήκη για τη Λειτουργία της Ένωσης. Και εφόσον Όλοι και όλες γνωρίζετε το περιεχόμενο του άρθρου 82. Θα ήθελα μόνο να σας υπενθυμίσω τις διατάξεις του άρθρου 3 της Συνθήκης Λειτουργία της Ένωσης. Τι λέει. Η Ένωση προσφέρει στους πολίτες της ένα χώρο ελευθερίας δικαιοσύνης και δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα όπου κατοχυρώνται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σε συνδυασμό με κατάλληλα μέτρα στον τομέα πρώτον ε, έλεγχο των συνόρων, άσυλο μετανάστευση και πρόληψη της εγκληματικότητας και καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Το άρθρο 3 λοιπόν αυτό συνιστά νέο στοιχείο που εισήγαγε η συνθήκη της Λισαβόνας Ο προκάτοχός του είναι το ε, παλιό άρθρο 2 της παλιάς συνθήκης όπου προσφέρεται ένας ε, χώρος ελευθερίας μέσω ενδεδειγμένων κατάλληλων μέτρων πρόληψης της εγκληματικότητας λέμε και καταπολέμησης του φαινομένου αυτού. Θα επανέλθω σε αυτό σε ένα λεπτάκι. Πριν όμως θα ήθελα να σας πω γιατί δεν συμφωνούμε γιατί δεν συμφωνεί η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου με την πρώτη σχολή, ενώ συμφωνεί εν μέρη με τη δεύτερη. Η πρώτη σχολή είναι, ε, ε, έχει έναν τρόπο ε, σκέψης περιοριστικό για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Γιατί βάσει αυτής της τάσης περιορίζεται η δυνατότητα έγκρισης της Ευρωπαϊκής Εντολής Προστασίας μόνο στις περιπτώσεις όπου υπήρξε ποινικό αδίκημα, το οποίο έχει εκδικαστεί ως ποινικό αδίκημα. Και βάσει των συζητήσεων που έχουν γίνει στι συναρμόδιε επιτροπές, ξέρουμε όμως ότι ο στόχος, και το υπενθύμησε και ο Πρόεδρος, ο στόχος είναι να προστατεύσουμε κάποιον κατά οποιοδήποτε κινδύνου. Άρα να περιορίσουμε την έκδοση της Ευρωπαϊκής Εντολής Προστασίας ε, μόνο όταν έχει κάποιος πέσει ήδη θύμα επίθεση ε, δεν διευκολύνει αυτό το άτομο. Δεν το επιτρέπουμε έτσι να κυκλοφορήσει ελεύθερα σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Έτσι συγχέεται η Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας με ένα προληπτικό μέτρο. Δηλαδή τι προλαμβάνουμε την επανάληψη της ε, αξιόπινης πράξης ε, και όχι όπως είναι ο εκπεφρασμένος στόχος της Ευρωπαϊκής Εντολής Προστασίας να προστατεύσουμε το άτομο πριν δεχτεί, πριν υποστεί την επίθεση. Η δεύτερη σχόλη τώρα της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου λέει ότι η νομική βάση άρθρο 82 δέλτα είναι καλή, αλλά προσθέτει και την μνήα στην ε, αμοιβαία αναγνώριση. Αλλά ε, παραμελεί το ότι θέλουμε να είναι ευρωπαϊκού χαρακτήρα το μέτρο αυτό, η Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Άρα δεν χρειάζεται η αναγνώριση των εθνικών αποφάσεων σε σχέση με ε, γιατί έτσι μπαίνουμε στο κανονικό καθεστώς αναγνώρισης αποφάσεων ή μέτρων, αν θέλετε, που έχουν αποφασιστεί σε ένα κράτος και πρέπει να αναγνωριστούν από το άλλο κράτος Όχι! Το ΕΠΟ είναι υπεράνω. Είναι ένα λεσέ πασέ επεκτείνει αυτόματα το εθνικό μέτρο. Οπότε το να προσθέσουμε ε, την, ε, το θέμα της αμοιβαία αναγνώρισης μας κάνει να καρκινοβατούμε σε σχέση με ε, την αυτοματοποίηση που, την έννοια της αυτόματης επέκτασης του εθνικού μέτρου που, μας, που κατοχυρώνεται με την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Τώρα, επανέρχομαι στη θέση μας, γιατί εμείς θεωρούμε ότι το 82-2 που διευκολύνει τη συνεργασία ανάμεσα στις δικαστικές ε, οι άλλες αντίστοιχες ε, αρχές συνιστά καλή βάση και ε, σε συνδυασμό βέβαια με το άρθρο 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε όλοι εδώ ότι η ευρωπαϊκές κοινότητες βασίστηκαν σε τέσσερις βασικές ελευθερίες, ε, κυκλοφορία των προσώπων, των αγαθών, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων. Μετά τη δεκαετία του 60 τι κάναμε, προσθέσαμε αυτό που τότε ονομάζαμε την πέμπτη ελευθερία κυκλοφορία των αποφάσεων και τότε είχαμε και τη σύμβαση των Βρυξελών για την αμοιβή αναγνώριση των αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Στο μεταξύ αυτό μετατράπηκε σε κανονισμό του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Εγώ θεωρώ ότι τώρα μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης Λισαβόνας έχουμε και έκτη ελευθερία η ελευθερία των πολιτών να κυκλοφορούν στο χώρο εμπλήρη ασφάλεια και δικαιοσύνη. Αυτή η ελευθερία περιγράφεται στο άρθρο 3. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει στους πολίτες της ε, την δυνατότητα να κυκλοφορούν ε, ελεύθερα σε έναν χώρο ασφάλειας και δικαιοσύνης μέσω ε, ενδεδειγμένων μέτρων ε, στον τομέα του ελέγχου αλλά και της ε, πρόληψης εγκληματικότητας και της καταπολέμησης αυτού του φαινομένου. Ξαναδιαβάζει ο μιλητής στο άρθρο 3. Γι' αυτό το λόγο και για τους πολιτικούς λόγους που επικαλέστηκε ο Πρόεδρος Εφόσον έχει την υποχρέωση να κατοχυρώσει αυτόν τον χώρο ελευθερίας και δικαιοσύνης η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αντιμέτωποι με ένα λίγαν ανησυχητικό φαινόμενο αυτό της ε, σεξουαλικής εγκληματικότητας, ας το πω έτσι, μέσα στις οικογενειακές αιστείες ε, ή σε ιδιωτικούς χώρους. Αντιμέτωποι λοιπόν με αυτό το φαινόμενο που έχει δυστυχώς ευρωπαϊκή διάσταση, πρέπει λοιπόν η Ένωση να κατοχυρώσει την προστασία. Προστασία, προστασία. Προστασία, έτσι, λέξη που χρησιμοποιώ. Δεν μιλάμε για πρόληψη. Το ποινικό δίκαιο ε, περιστρέφεται γύρω από αυτήν την έννοια του επικίνδυνου, της επικίνδυνης συμπεριφοράς του ατόμου κατά της οποίας πρέπει να προστατεύσουμε το, το ιονή θύμα. Ε, ε, μια, αν μια γυναίκα προστατεύεται ήδη στο κράτος μέλος όπου διαμένει, θα πρέπει να, η προστασία να τη συνοδεύσει εκεί όπου θα πάει μέσα στα πλαίσια του χώρου ελευθερίας και δικαιοσύνης. Και για να γίνει αυτό, για να τύχει αυτή τη προστασία, πρέπει να επεκτείνουμε την προστασία στο άλλο κράτο μέλο που θα πάει να ζήσει αυτή η γυναίκα. Αυτή η επέκταση τη προστασία γίνεται μέσω τη ε, υιοθέτηση ε, τη Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασία που δεν χρειάζεται να αναγνωριστεί από το άλλο κράτο μέλο αυτόματα. Επεκτείνεται υπό την προπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτούμενοι όροι για να εκτελεστεί στο άλλο κράτο μέλο. Γιατί οι αρχέ, άσχετα με το αν είναι δικαστικέ, αστικέ, ποινικέ, διοικητικέ, πολιτικές, αυτές οι αρχές πρέπει να βασίζονται ε, στην αρχή που σαφέστατα προσδιορίσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mutual trust, αμοιβαία εμπιστοσύνη. Εάν μια δικαστική αρχή ε, ενό κράτου μέλου έχει εκδώσει μέτρο προστασία, ε, πρέπει εγώ να εμπιστευτώ, εγώ ποιο είμαι, η αρχή ενό άλλου κράτου μέλου, πρέπει να εμπιστευτώ την αρχή του πρώτου κράτου μέλου και να ε, εγγυηθώ την προστασία αυτού του ατόμου. Γι' αυτό με στη δική μας γνωμοδότηση, τη γραπτή μου γνωμοδότηση, επιβεβαιώνουμε ότι η νομική βάση αυτής της οδηγίας είναι όντω το άρθρο 82 πρώτη παράγραφος εδάφιο δέλτα σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ένωσης. Εν κατακλείδη, Α, μπορεί να μας πει κάποιος, μα υπάρχουν δύο ε, ε, δύο διαφορετικές συνθήκες, γιατί το 82 είναι στη συνθήκη για τη λειτουργία και το άλλο, το άρθρο 3, είναι στη συνθήκη της Ένωσης. Λοιπόν, σήμερα μετά την ε, θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, ε, οι δύο συνθήκες ε, συνιστούν ένα ενιαίο έρισμα επί το οποίο δράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση το ότι έχουμε μία νομική βάση σε μία συνθήκη και μία άλλη στην άλλη συνθήκη δεν συνιστά νομικό μειονέκτημα για την έγκριση της οδηγίας. Θα κλείσω την παρέμβασή μου και θα μείνω στην διάθεσή σας αν τυχόν έχετε ερωτήματα και σας ευχαριστώ για την προσοχή που δείξατε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. ακούγοντας την ε, εξαντλητική αυτή και αναλυτική ε, παρουσίαση της νομικής υπηρεσίας έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε τους συνεισηγητές της Επιτροπής μας και της Επιτροπής Γυναικών. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Ρομέρο Λόπες που είναι η συγγήτρια της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα με γνήσιο ενδιαφέρον τη νομική ε, υπηρεσία του Κοινοβουλίου και τη γνωμοδότησή της και επειδή η πρωτοβουλία αυτή ήταν αγώνας ε, δρόμου με τεμποδίων μέχρι να φτάσουμε σήμερα ε, στην παρουσίαση της έκθεσής μας Πρέπει να σας πω ότι ευχαριστώ τη Γραμματεία και τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου γιατί πραγματικά τερματίσαμε αυτόν τον αγώνα με το εμποδίο. και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν εκεί και τους συνεργάτες μας και τους βοηθούς μας και των δύο εισηγητών και αυτό είναι επίση μια καινοτομία. Συμμετέχουν δύο επιτροπές ε, στην υπόθεση αυτή η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου στη γνωμοδότησή της βάζει μια νέα φιλοσοφία στην πρόληψη της ε, εγκληματικής πράξης και την προστασία του θύματος. Ε, είναι λοιπόν ένα μέτρο ασφαλιστικό εκ των προτέρων πριν την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων. Και εδώ λοιπόν έχουμε ένα ε, στοιχείο νεοτερισμού πώς να το πω, με πραγματικό αντίκτυπο. Σε πρώτη ανάγνωση εκρίθηκε έτσι. Το 1985 ε, ήδη ρυθμίστηκε αυτό το θέμα και της προστασίας των ε, θυμάτων και το 2001 σε απόφαση πλαίσιο και το 2009 σε οδηγία. Γίνεται λόγος για το καθεστώς του θύματος και του συστήματος ε, αποζημίωσης, αλλά δεν μιλάει κανείς για την πρόληψη της τέλεσης αξιόπινης πράξης. Κάτι άλλο που θα ήθελα να τονίσω είναι το εξή. Δεν είναι μόνο το άρθρο 3 της Συνθήκης Λισαβόνας που τόσο καλά εξήγησε ε, η νομική υπηρεσία, αλλά και ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων που επισυνάπτεται στο ε, κείμενο της συνθήκης και είναι βασικό κείμενο για τις αξίες και στο πρώτο τίτλο ορίζει ότι τα βασανιστήρια, η κακοποίηση, η δολοφονία, η ανθρωποκτονία κτλ μπορεί να είναι από ένα πολύ κοντινό πρόσωπο του θύματος και πολλές φορές από την ίδια την οικογένεια. Ο τίτλος πρώτος λοιπόν μιλάει για την αξιοπρέπεια ε, του ατόμου απέναντι ε, ε, στην βία και θα πρέπει αυτός να προστατεύεται το θύμα από μια κρατική αρχή. Λοιπόν, εδώ δεν νοείται ε, ιδιωτική σφαίρα. Ό,τι είναι προσωπικό είναι και πολιτικό. Δεν υπάρχει προσωπική ιδιωτική βία, είναι κρατική βία. Και θα πρέπει το κράτο να προστατεύει και να κάνει πραγματικότητα αυτή την πρωτοβουλία. Δεν είναι πρωτοβουλία δύο κρατών μελών αυτή, προσέξτε. Δεν είναι πρωτοβουλία τη Ισπανική Προεδρία. Αλλά ε, χιλιάδε γυναίκε το ζητούν αυτό και όχι μόνο γυναίκε και άλλα θύματα. Wave που είναι ε, μια μη κυβερνητική οργάνωση ε, ομιλεί για 2.500 γυναίκες που έχουν δολοφονηθεί στην Ευρώπη και είναι τα στοιχεία ακόμα άγνωστη. Στην Ισπανία εκκρεμούν 118.000 παρακαλώ εντάλματα προστασίας και φέτος ε, μπορεί άλλα 40.000 ε, να προσθεθούν. Και στην Ευρώπη, την υπόλοιπη πάλι 100.000. Όλα αυτά είναι στοιχεία ε, κατά προσέγγιση και δεν μπορούν να ε, γίνουν γενικέ προβολέ, αλλά τι κάνουμε μοιραία γιατί δεν έχουμε όλα τα στοιχεία στα χέρια μα. Ακούστηκαν και ε, επιχειρήματα κατά της προσπάθειας αυτή, ότι το θύμα θυματοποιείται για δεύτερη φορά, ότι επιδοτούμε δικηγόρου, ότι γεννάμε φρούδες ελπίδες, ότι όλα αυτά είναι προκαταλήψεις. Πολλέ φορές είναι και άγνοια όμως, γιατί ε, ε, δεν καταλαβαίνουν αυτοί που τα λέγουν αυτά την έννοια του κειμένου, το πνεύμα του κειμένου. Στα χέρια μας είναι να πετύχει αυτή η προσπάθεια και να γίνει μια μελέτη αντικτύπου για να δούμε πού υπάρχουν προβλήματα, πού υπάρχουν δυσκολίες, οποία στραγγαλίζεται το κείμενο. Εμείς δεν θέλουμε να στραφούμε κατά των διαφόρων ε, νομικών πολιτισμών ή παραδόσεων. θέλουμε να βοηθήσουμε, να συνεργαστούν. Και ακόμα και, ένα, και μόνο θύμα να βοηθήσουμε, πραγματικά θα άξιζε τον κόπο. Οποιαδήποτε πρωτοβουλία βελτιώνει αυτό που σήμερα συζητούμε, θα πρέπει να λάβει υπόψη της την ευρωπαϊκή περιπλοκότητα. Θα πρέπει να λάβει υπόψη της τις νομικές μας παραδόσεις και τις διαφορές τους. Ας μην αρχίσουμε όμως να ε, μειώνουμε και να την κατηγορούμε και να πούμε ότι θα αποτύχει, θα είναι αποτελεσματική. Όχι, να φροντίσουμε να είναι αποτελεσματική. Και γι' αυτό καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον να σκεφτεί τη θέση της, να την αναθεωρήσει για να μπορέσει αυτή η προσπάθεια να ευδοκιμήσει. Και στο μέλλον να έχουμε καλύτερη προσέγγιση των ε, κρατών μας. Μερικά σημεία έχουν διαγραφεί από το κείμενο του Ιανουαρίου και θέλουμε να τα επαναφέρουμε για να βελτιώσουμε ή να διευκρινίσουμε ορισμένε καταστάσεις ε, που αντιμετωπίζουν τα θύματα. Ε, επίσης όμως είναι σημαντικό κατά την άποψή μα να επιμείνουμε στην πρόληψη Λοιπόν, δεν είναι άλλο ένα κείμενο. Όχι, τώρα αρχίζει αυτή η προσπάθεια. Ε, τώρα ε, αρχίζει η πραγματική πορεία με τις προτάσεις των διαφόρων ε, βουλευτών από τις διάφορες πολιτικές ομάδες για να βελτιωθεί η πρόταση και να ε, επιτευχθεί και ο στόχος της άλλωστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Ρομέρο. Και τώρα για να ολοκληρώσουμε με την παρουσίαση της πρότασης θα ακούσουμε τη συνεισηγήτρια, την κυρία Χιμένεθ Πεθερίλ, από την Επιτροπή Γυναικών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τη νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου, διότι αντέδρασε ταχύτητα. Δεν ήξερα καν ότι σήμερα θα μας παρουσίαζαν την γνωμοδότησή τους, αλλά τους ευχαριστώ ιδιαιτέρως, διότι ρίχτηκε φως αυτή την υπόθεση εντολής προστασίας και συμφωνώ μαζί τους όταν μιλάμε για προστασία. Η προστασία του θύματος είναι αυτή που είναι πιο σημαντική. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Ρομέρο η συγγήτρια σε αυτή την κοινή πρωτοβουλία, καθώς επίσης και τη γραμματεία της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, της Επιτροπής ΦΑΜ και όλους όσους ε, συμμετείχαν ε, για αυτή την, σε αυτή την τόσο δύσκολη έκθεση, διότι λάβαμε πάρα πολλές εκδοχές από το Συμβούλιο, οι οποίες έκαναν ουσιαστικές αλλαγές στο αρχικό κείμενο και εμείς χρειάστηκε να προσαρμοζόμαστε συνεχώς και όλα αυτά σε χρόνο ρεκόρ, διότι υπάρχει αυτή η πίεση χρόνου για να έχουμε ε, ψηφοφορία προσανατολισμού εντός του Ιουνίου. από αυτό που ακούσαμε καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλέ ελπίδε. Διότι γνωρίζουμε ήδη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πει και δημοσίω αλλά και κατηδίαν στι ε, συνεδριάσει εργασία που είχαμε τι αμφιβολίε τη για την νομιμότητα αυτή τη πρωτοβουλία. Στη συνεδρίαση που είχαμε την περασμένη Τρίτη μεταξύ εμπειρογνωμένων ε, οι οποίοι συζήτησαν τα πιο διαφιλονικούμενα θέματα σε αυτή την αξιολόγηση αντικτύπου, προέκυψε το θέμα των ε, διαφορετικών ε, νομικών βάσεων για την εφαρμογή, διότι ανάλογα με τη χώρα υπάρχει διαφορετική ε, μεταχείριση και άλλες φορές είναι ποινική και άλλες φορές είναι διοικητική η ποινή. Δεν θα επισέλθω εγώ σε λεπτομέρειες, ακούσαμε την νομική υπηρεσία του Συμβουλίου και εγώ θα ήθελα σήμερα να μας πει και την άποψή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ρίξουμε περισσότερο φως στην υπόθεση. Αυτό που διαπιστώνω είναι ότι τόσο το Συμβούλιο όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούν να βρουν λύσεις για να έχουμε πρακτική εφαρμογή αυτού που προσπαθούμε να επιτύχουμε όλοι, προστασία των θυμάτων. Το Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα να ε, βελτιώσει αυτή την πρωτοβουλία, αλλά χρειαζόμαστε ένα πραγματικό πλαίσιο της πραγματικής κατάστασης αυτή τη στιγμή. Τα κράτη-μέλη που την υποστηρίζουν, τη νομική βάση, την οποία αυτή τη στιγμή διευκρινίζουμε και την αποτελεσματικότητα του μέτρου αυτού. Ελπίζω το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώσουν το συμμετομότερο δυνατόν για να μπορέσουμε να εργαστούμε καλύτερα στο μέλλον με την έκθεση αυτή. Ως εισηγήτρια, εγώ έλαμβανα υπόψη το αρχικό κείμενο που μας είχε δώσει το Συμβούλιο και οι τροπολογίες μου έγιναν προς αυτό το κείμενο. Επειδή το τελικό κείμενο θα το έχουμε στις 4 Ιουνίου μεταξύ άλλων, τότε θα προσθέσουμε και περισσότερες τροπολογίες ε, σε αυτό το οριστικό κείμενο. Παρόλα αυτά, και παρά το γεγονό ότι η εξέλιξη αυτή τη έκθεση, όπω είπε η κυρία Ρομέρο και επαναλαμβάνω εγώ, δεν ήταν ένα δρόμο σπαρμένο με ρόδα, εγώ εξακολουθώ να επιμένω διότι η προστασία των θυμάτων που είναι αυτό το οποίο προσπίζομαι εγώ εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, διαπιστώνω είναι ότι, ότι είναι αυτό που ξεχνούμε κάθε φορά. Και κάθε φορά που υπάρχει δυνατότητα, εγώ υψώνω τη φωνή μου ώστε να καλύπτεται αυτό το θέμα της προστασίας των θυμάτων. Κυρίως ε, θύματα γυναίκες που ορισμένες φορές ε, λαμβάνουν εντολή προστασίας και θέλουν να μετακινηθούν εντός της Ευρώπης. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι όταν θέλουμε να προστατεύσουμε τα θύματα και θα πρέπει να σκεφτόμαστε και όλες τις γυναίκες οι οποίες είναι θύματα ε, υποχρεωτικών γάμων, ε, εμπορίας ανθρώπων, οργανωμένου εγκλήματος, θύματα τρομοκρατίας ε, και αυτό φέρεται και στην ε, τροπολογία μου υπαριθμών 6. Επίσης θέλησα να επισημάνω την προστασία της αξιοπρέπειας του θύματος, διότι δυστυχώς γνωρίζω πάρα πολύ καλά το σύμπαν του θύματος, διότι όπως θα γνωρίζετε, ε, η ΕΤΑ σκότωσε τον αδερφό μου και τη γυναίκα του και Ξέρω από ίδια πείρα ότι όλοι όσοι βρίσκονται στην κατάσταση του θύματος πρέπει να προστατεύονται και πρέπει να προστατεύεται και η αξιοπρέπειά τους. Επίσης με ενδιαφέρει και η προστασία των ανηλίκων, ε, διότι μπορεί να βρεθούν ενώ, ε, ε, εντός μιας οικογενειακής διαμάχης. Και είναι πολύ σημαντικό επίσης να μην δρούμε μόνο κατά ενός ανθρώπου, αλλά και ομάδων που μπορεί να αποτελούν απειλή για το θύμα. Αυτό είναι η τροπολογία 27. Και επίσης ε, η προστασία του θύματος και για να μπορέσουμε ε, να αναγνωρίζεται η εντολή, διότι ορισμένες φορές μπορεί να αναγνωρίζεται, ε, θέλω να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ε, δεν αναγνωρίζεται μια εντολή, διότι αλλιώς δεν μπορούμε να, να αναζητήσουμε λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν από αυτή τη, αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να έχουμε συνένεση. Εγώ σκέφτομαι στο θύμα, στο οποίο θα πρέπει να υπάρχει ε, μια εξασφάλιση νομική και είτε θέλει να μετακινηθεί σε μια χώρα είτε θέλει να περιμείνει στη χώρα του. Γι' αυτό λοιπόν σε περίπτωση που δεν αναγνωρίζεται η εντολή προστασίας θα πρέπει να ενημερώνεται το θύμα. Αυτό είναι στο άρθρο 29, το οποίο κατά την άποψή μου είναι διαφιλονικούμενο, διότι αυτή η εντολή θέλει να διευκολύνει τη ζωή του θύματος. Και αν το θύμα πρέπει να ξεκινήσει μια νέα διαδικασία για να λάβει μια νέα εντολή προστασία στη χώρα στην οποία θα μετικήσει, χάνεται όλη η αξία αυτής της εντολής. Αυτό ανέφερε και ο εκπρόσωπος ε, της νομικής υπηρεσίας ε, και είπε ότι θα πρέπει να γίνεται αυτομάτως. Η τροπολογία και η αιτιολογική μου έκθεση έχουν ένα στόχο. Το θύμα να μην πρέπει να ξαναμπεί στη νέα διαδικασία αναζήτησης μια νέα εντολής. Ε, στη, ξένη, στη χώρα μου μόνο ένα 8% κάνει καταγγελία για να λάβει μια τέτοια εντολή προστασίας. Φαντάζεστε τι θα γίνεται αν αυτοί οι άνθρωποι φτάσουν να μετικήσουν σε μια ξένη χώρα. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την παράγραφο 2 του άρθρου 2 που λέει πώς μπορούμε να προστατεύσουμε πραγματικά έναν άνθρωπο που χρειάζεται ανάγκη προστασίας, εντολή για να ε, μην πλησιάζει κάποιο την προσωπική του κατοικία και άλλα μέτρα τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται σε όλες τις χώρες η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει πόρου προκειμένου να προστατεύει οργανώσει που προστατεύουν τα θύματα, ε, οργανώσει οι μπορούν να πάνε τα θύματα για να λάβουν πληροφορίε για το τι ακριβώ μπορούν να κάνουν για την κατάστασή του. Θα πρέπει να υπάρχει ηθική προστασία εντό αυτών των οργανώσεων, εάν ε, την χρειάζεται το θύμα και αυτή είναι η τροπολογία μου υπαριθμών 9. Οι τροπολογίε μου προσπαθούν να προστατεύσουν όλα τα θέματα και ε, θύματα και λέω όλα τα θύματα, διότι όταν μιλάμε για προστασία Μιλάμε για συμπεριφορές οι οποίες μπορεί να μην είναι ποινικές, ε, ποινικά κολάσιμες, αλλά μπορεί να οδηγηθούν σε ε, τέτοιες συμπεριφορές. Μπορεί να έχουμε απειλές οι οποίες μπορεί να δυσχεραίνουν τη ζωή ενός ανθρώπου. Αυτό αναφέρεται και στην τροπολογία μου 24. Στην αιτιολογική έκθεση ε, βλέπετε τα στοιχεία τα οποία έχουμε προσθέσει ως συνεισηγήτρες στο κείμενο του Συμβουλίου θα πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ ότι έχουμε ε, ένα πολύ καλό μέσο το οποίο θα μπορούσε να μας οδηγήσει να προστατεύουμε ουσιαστικά τα θύματα αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να λύσουμε και τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από την εντολή αυτή προστασίας και τα οποία Μα επισυνώνονται από διάφορε οργανώσει, όπω για παράδειγμα τη Βρετανική Οργάνωση Justice, η οποία θεωρεί ότι αυτή η πρωτοβουλία θα πρέπει να γίνει ε, κοινή συνενέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το European Women Lobby, το οποίο εκφράζει κάποιε ανησυχίε για τις ε, διακρίσει που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ θυμάτων από διάφορε χώρε. Θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι, να ξεχνούμε προσωπικά συμφέροντα, είτε συμφέροντα χώρα, συζητητή ή θεσμικού οργάνου, διότι το θύμα είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να έχει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο ώστε να είναι προστατευμένο στι 27 χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Και επίση αυτό θα πρέπει να γίνεται ταχύτατα και αποτελεσματικά και να μην πρέπει τα θύματα να ξεκινούν νέε δικαστικέ διαμάχε επειδή υπάρχει διαφορά ε, στην ε, νομοθεσία και την ομολογία των διαφόρων κρατών μελών. Θα πρέπει να βρούμε λύσει υπεύθυνε και το να προσπαθούμε να έχουμε ε, ταχεία επιτυχία να μην αποτελέσει τροχοπέδι στην ε, ε, εξέβρεση λύσης για το θέμα μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που μας βοηθούν να εμπληκτούσουμε το κείμενο αυτό για την οδηγία αυτό, αυτή και επίσης θεωρώ ότι το θέμα της προστασίας των θυμάτων, όπως αναφέρεται και στο πρόγραμμα της ε, Στοχόλμης, ε, θα πρέπει να είναι μία από τις επιτυχίες αυτής της θητείας και θα πρέπει να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε σε ένα χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας. Ευχαριστώ. Τα μέλη των Επιτροπών τώρα, ε, Ελευθεριών και Γυναικών, αλλά προηγουμένως θα πρότεινα να ακούσουμε την Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ σύντομα, διότι ε, είναι κοινή η συνεδρίαση και σίγουρα έχουν και άλλες ανηλυμένες υποχρεώσεις τα μέλη των δύο επιτροπών. Παρακαλώ. Να ακούσουμε πρώτα την Προεδρία και μετά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια τους βουλευτές των δύο επιτροπών μας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε της Επιτροπής Γυναικών. Σας ευχαριστώ και πάλι που μας δίνετε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να παρευρισκόμαστε για να συζητήσουμε την πρωτοβουλία αυτή, όπου όπως πολύ καλά είπατε είναι πρωτοβουλία 12 κρατών μελών. Δεν είναι ισπανική πρωτοβουλία, είναι 12 τα κράτη-μέλη, διότι όλοι οι εμπνευστές όλοι ανεξαιρέτως υποστήριξαν ε, εξόχως την πρωτοβουλία αυτή. Και δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερους ε, εμπνευστές, επαναλαμβάνω, γιατί η υποστήριξη των κρατών μελών ήταν πάντα άριστη. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων προσθέθησαν και άλλες χώρες που υποστήριξαν ε, με τεπιτάσεως αυτά τα θέματα και είμαστε πολύ περισσότεροι από 12. Δεν ξέρω πόσοι. Στις 4 Ιουνίου θα το διαπιστώσουμε αυτό στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης. Θα πρέπει βεβαίως να ευχαριστήσουμε την νομική υπηρεσία ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εργασία του για την πρωτοβουλία αυτή, διότι όπως πολύ σωστά είπε είναι καινοτόμα και ρηξικέλευθη. Και στην αρχή ο κόσμος φοβάται οτιδήποτε το νέο και το πρωτοφανές και, και στη συνέχεια αισθάνεται ανασφάλεια. Ε, νομίζω όμως ότι η νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διασκέδασε απολύτως το φόβο και μας καθησύχασε όλους. Και μάλιστα σε έναν χρόνο ρεκόρ. Διότι καταλαβαίνουμε ότι το θέμα είναι πάρα πάρα πολύ περίπλοκο και ειλικρινά το να εκδώσει κανείς ε, κατευθυντήριες γραμμές τόσο σύντομα μας ε, φαίνεται ειλικρινά εξαιρετικό, θαυμάσιο και ευχαριστούμε ε, τη νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου για την καλή δουλειά ε, σε αυτή την υπόθεση. Και βεβαίως συμφωνούμε με τα επιχειρήματά σας ε, για τη νομική βάση. Υπό την έννοια αυτή δεν υπάρχει καμία ε, διχογνωμία στο Συμβούλιο και βεβαίως γνωρίζουμε και συμφωνούμε ότι στόχος είναι, όπως πολύ ωραία υπογράμμισε η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου, είναι η προστασία. Για την έκθεση την ίδια θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, Πρόεδρε. η κοινή έκθεση της Επιτροπής Γυναικών και της Επιτροπής ε, Ελευθεριών ε, είναι μια προσπάθεια που θα χαρακτηρίζαμε ως εξής από την Προεδρία. Ε, είναι θαυμάσια και λαμπρή προσπάθεια που προχωρεί προς μια κατεύθυνση πολύ καλή, πολύ φιλόδοξη, έχει πολλά στοιχεία, επίσης καινοτόμα, γίνεται λόγος για στατιστικές εδώ και δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει στατιστικές. Σήμερα δεν έχουμε στατιστικές, δεν μπορούμε να τις συγκρίνουμε. Γι' αυτό μιλάει η έκθεση. Επίσης ε, μιλάει για την πρόληψη, για τις ενημερωτικές εκστρατείες που είναι πάρα πολύ θεμελιώδη στοιχείο και αυτό για να επιτύχουμε πραγματική προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ένα τρίτο στοιχείο που θα ήθελα να υπογραμμίσω εδώ γίνεται λόγος για την αξιοπρέπεια του θύματος. Διότι το θύμα πραγματικά αυτό που ζητάει δεν είναι αποζημίωση χρηματική. Θέλει να γίνεται σεβαστή η αξιοπρέπειά του. Αυτό ζητάει και ε, κάποια προστασία και υποθέση. Ε, υπόθαλψη. Ευχαριστούμε τη νομική υπηρεσία και βεβαίως τις δύο εισηγήτριες για την εξαιρετική τους εργασία και τους συνεργάτες και τους βοηθούς. Ξέρω ότι ήταν δύσκολη η προσπάθεια αυτή για όλους, αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα που έχουμε ενώπιόν μας είναι απλούστατα ε, πολύ ελπιδοφόρο και φιλόδοξο και στο λίγο χρόνο που μένει στην Ισπανική Προεδρία ε, θα ε, δώσει συνέχεια ε, στην προσπάθεια αυτή και θα συνεργαστεί και με το Βέλγιο που θα μας διαδειχθεί όπως και το Βέλγιο συνεργάστηκε μαζί μας. Ευχαριστώ κύριε Μολίνος. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάλι σύντομα σας παρακαλώ να ακούσουμε τον κύριο Αλτάν ή τον κύριο Σόνσκα, δεν ξέρω ποιος είναι εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you, Mr. Chairman. And thank... Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε για τις παρουσιάσεις και για τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας ε, προσβλέπουμε με υπομονησία σε αυτή την γραπτή γνωμοδότηση. Θέλουμε να την αναλύσουμε. Ανέκαθεν ναι, υποστηρίζαμε τους στόχους αυτής της πρωτοβουλίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό αληθεύει ακόμη και σήμερα. Έχει θέσει ω ύψιστη προτεραιότητα την προστασία των θυμάτων, την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξετάζουμε αυτά τα ζητήματα τώρα, διότι διεξάγουμε και αξιολόγηση αντικτύπου ε, για να δούμε με ποιο τρόπο θα μεριμνήσουμε ώστε να κατοχυρώνονται τα δικαιώματα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Το 2011 θα υποβάλουμε νέα πρόταση, ένα ευρύ φάσμα και μέσα σε αυτή την ανάλυση θέλουμε να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο και το Συμβουλίο για να βρεθούν λύσεις σε οσδήποτε δυσκολίες ανακύψουν. Σημαντικά ζητήματα, όπως ανέφεραν οι συνάδελφοι, είναι ε, η ενημέρωση, ε, η ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης των θυμάτων. Όλα τα θέματα αυτά θα τα αναλύσουμε και στο εγγύς μέλλον θα σας υποβάλουμε μία πρόταση. Αναφέρθηκε ο συνάδελφος ε, στην συνεδρίαση εμπειρογνωμών την περασμένη εβδομάδα. Μπορούμε να σε ενημερώσουμε για την έκβαση της συνεδρίασης, αν σας ενδιαφέρει. Αν το χρειάζεται, ζητήστε το. Είπα ότι αυτό το θέμα είναι ύψη της προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να βρούμε ε, λύσεις κατάλληλες σε σχέση με την ε, νομική βάση που έχει προσδιοριστεί. Ευχαριστούμε κυρία Άλτον. Τώρα θα ακούσουμε τα μέλη της Επιτροπής. Περιορίστε το χρόνο αγόρευσή σας, ε, παρακαλώ, για να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη των δύο επιτροπών γίνεται, γιατί δεν έχουν ε, όλοι την, τις ίδιες ε, απόψεις. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες υποχρεώσεις. Thank you very much indeed, President. Uh, <clears throat> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι ορόσημο αυτή η έκθεση. Είναι σημαντικό γιατί δείχνει σε ποιο τομέα υπάρχουν ανησυχίες στο Κοινοβούλιο. Ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ε, ε, μέτρο σύγκρισης, αν θέλετε, αυτό το σχέδιο. Θα μιλήσω με την ιδιότητα του νομικού και επειδή έχω και εμπειρία στον τομέα του οικογενειακού δικαίου και της οικογενειακής βίας. Ανησυχώ ε, και για τη νομική βάση και για τις επιπλοκές που ενδέχεται να ανακύψουν αν εγκριθεί η Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Προβλήματα και διλήμματα προκύπτουν από τις διαφορές στα ένωμα συστήματα των κρατών μελών, ε, η φύση της βίας, πώς αντιμετωπίζεται στα επιμέρους κράτη σχέση ανάμεσα στο αστικό και ποινικό δίκαιο και σε κάθε περίπτωση η εφαρμοσιμότητα αυτού του ε, συστήματος μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες, σε περιπλοκές. Ο απότερος στόχος και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε είναι να υπάρχει καταδίκη πριν εκδοθεί η εντολή. Οπωσδήποτε. να το να έχουμε ένα ομιχλώδες ε, σύστημα, μια σαφή προσέγγιση δεν είναι το ευκταίο, γιατί από νομική σκοπιά, το ξέρετε, ε, όταν είναι ασαφής ε, η κατάσταση μπορεί κάποιοι να εκμεταλλευτούν τις διατάξεις με δόλιες προθέσεις. Για την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων θέλω ορισμό γι' αυτό. Εξέτασα προσεκτικά τα ζητήματα. Όλοι είμαστε ιονοί θύματα. Η προσέγγιση μηδενικής ανοχής ε, είναι πολύ δύσκολη. Φυσικά για την ευεία κατά των γυναικών, ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την προσέγγιση χρειαζόμαστε. Αλλά τώρα να τα βάλουμε όλα τα στο ίδιο σακούλι, όλες τις πιθανές και αληθινές ε, αξιόπινες πράξεις να τις ε, ομαδοποιήσουμε σε μια τέτοια αντικειμενική προσέγγιση και με μια ευρωπαϊκή εντολή προστασίας είναι κάτι το ανέφικτο κατά τη γνώμη μου. Ειλικρινά συμφωνούμε για κάποια σημεία. Τροπολογία 10 παραδείγματο χάρη. Ε, είναι πολύ σημαντικό να ισχύει το ένομο να προσαρμοστεί το ένομο σύστημα κάθε κράτους μέλους και στις διατάξεις της νομικής βάσης προβλέπεται αυτό, δηλαδή να προσαρμοστεί το σύστημα στην Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας, να ε, υπάρχουν σαφή όρια. Τροπολογία 66 επίσης, εκεί εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με τα ε, μέτρα ε, στέρησης της προσεπικής ελευθερίας που αναιρούν Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας, αν αυτή έχει βασιστεί σε δικαστική απόφαση. Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί λοιπόν να ασχοληθεί με τέτοια μέτρα, custodial measures, μέτρα στερητικά της προσωπικής ελευθερίας. Τι εννοούμε και χρειάζεται δικαστική απόφαση, είτε είναι στο πλαίσιο του ποινικού δικαίου καταδίκη, είτε αστική απόφαση σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά εδώ λέμε τα αντίθετα. Ε, και άρα είναι ε, χωλένη η πρόταση. Λοιπόν, είναι καλό μετροσύγκριση στο σχέδιο, αλλά από πλευράς νομικής ε, βάσης δεν επαρκεί. Ε, η πρόταση. Δεν είναι εφικτό τον ε, να επιτύχουμε τους στόχους μας αν επικρατήσει ένα ομιχλώδες νομικό ε, τοπίο. Δεν θα προστατεύσουμε έτσι τις γυναίκες και τα δικαιώματά τους και οτιδήποτε κάνουμε εδώ πέρα μπορούμε να με οτιδήποτε κάνουμε μπορούμε να προστατεύσουμε όσους κινδυνεύουν. Η Νάταλη Γκρίσπεκ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομη. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Ευχαριστώ τους ε, εισηγητές και τα επιτελεία τους για την ε, πρόοδο που έχει σημειωθεί, γιατί είναι εξαιρετικά περίπλοκο το σχέδιο, το προανέφεραν οι συνάδελφοι. Ε, θα ήθελα να πω πως ε, στο οικοδόμημα, στην οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουμε ένα συγκεκριμένο βήμα με την έγκριση και την έγκριση των τροπολογιών αυτού, για αυτό το σχέδιο. Αυτή η πρωτοβουλία συνιστά ε, πρόοδο, το είπαν οι συνάδελφοι, δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί κανείς άκουσα τις απόψεις ε, των εμπλεκόμενων. Ευχαριστώ την νομική υπηρεσία ε, που μας διαφώτισε για το περιεχόμενο αυτού του σχεδίου που καλούμε θα να εγκρίνουμε. Είναι περίπλοκο το θέμα, είναι περίπλοκο το ζήτημα της νομικής βάσης, αλλά δεν είναι και ακριβής επιστήμη. Το δίκαιο το ξέρουμε όλοι, πλην όμως ε, ή μάλλον είναι θέμα ερμηνείας των διαφόρων νομικών ε, υποσημείων. Οι δύο επιτροπές, Επιτροπή Λίμπε και Επιτροπή Γυναικών, εργάστηκαν σκληρά για το σχέδιο και αποτελεί καινοτομία στην εργασία τους. Άλλη καινοτομία είναι το, το, το περιεχόμενο, δηλαδή η προστασία των θυμάτων, των ιονή θυμάτων. Αυτό είναι σχεδόν επαναστατικό. Η ιδέα της επέκτασης της προστασίας που ανέφερε η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου, η επέκταση του μέτρου είναι κάτι το επαναστατικό. Αν περάσει αυτή η πρόταση θα ε, πραγματοθεί το περιεχόμενο του άρθρου 3 σε Ευρωπαϊκή Ένωσης. Δηλαδή θα κυκλοφορούμε ελεύθερα, ε, ελευθερία, δικαιοσύνη. Και όχι μόνο αυτό. Θα υπάρχει ε, νοσιακή προστασία Δηλαδή θα επεκταθεί η εθνική προστασία και θα γίνει η ευρωπαϊκή προστασία. Είναι καταπληκτικό. Εν κατακλείδη. Με τη συνδρομή όλων μας θα προχωρήσει αυτή η πρόταση. Η δε πρακτική εφαρμογή αυτής της νομικής πράξης ε, θα συναντήσει δυσκολίες. Σίγουρα θα είναι περίπλοκο, αλλά σίγουρα θα είναι και δύσκολο να εφαρμοστεί ε, η πράξη αυτή, αλλά πάντως έτσι κάνουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα μέσα στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα γιατί μεταφράζουμε στην πράξη τα περιεχόμενα της συνθήκης της με την ε, ε, κοινή συνεργασία των δύο επιτροπών. κυρία Ντελήλ. Η κυρία Ντζελίλη, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει χρόνος για να μπορέσουμε να κάνουμε τις κατάλληλες διορθώσεις ώστε να επισημάνουμε τα κατάλληλα στοιχεία, ώστε το κείμενο να είναι το καλύτερο δυνατόν και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα δικαιώματα των θυμάτων. Θα ήθελα πραγματικά σήμερα να ευχαριστήσω τις δύο συνεισηγήτριες. Συμφωνώ απολύτως με τη γνωμοδότησή τους ε, και με τα στοιχεία τα οποία έχουν προσθέσει στη συζήτηση. Γι' αυτό δεν θα ήθελα να επισέλθω σε θέματα ουσίας, δεν θα ήθελα να επαναλάβω τα ίδια στοιχεία τα οποία μας είπαν οι συνεισηγήτριες. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να τονίσουμε την άποψη της νομικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία μας εδόθη, και να επισημάνουμε ότι κατά κάποιο τρόπο είναι επαναστατική. Ίσως το επαναστατική είναι υπερβολικό, αλλά νομίζω ότι αυτή η γνωμοδότηση είναι σημαντική, διότι η νομική υπηρεσία μας είπε και θέλησε να λάβει υπόψη του το ναι, ένταλή αυτή προστασίας όχι ως απλό προληπτικό μέτρο, ένα μέτρο το οποίο θα είναι συμπληρωματικό, επικουρικό και το οποίο μπορεί να αναγνωρίζεται μεν σε ένα κράτος μέλος, αλλά σε κάποιο άλλο μπορεί να μην αναγνωρίζεται ή να αναγνωρίζεται με διαφορετικό τρόπο. Η νομική υπηρεσία θέλησε να τονίσει ότι η εντολή προστασίας είναι δικαίωμα στην προστασία και σημαίνει αυτό ότι είναι αναπόσπαστο τμήμα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των δικαιωμάτων του θύματος. Επομένως, αν αντιληφθούμε έτσι την εντολή προστασίας, ενισχύονται τα δικαιώματα των θυμάτων και εγώ θα έλεγα τα δικαιώματα των ανθρώπων και φυσικά ενισχύεται και η ε, σαφήνεια της ποινή. Επίσης, δεν θα πρέπει να περιοριστούμε απλώς και μόνο στην αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων βάσει της νομικής ε, βάσης, αλλά θα πρέπει, δεδομένου ότι το κύριο σημείο αναφοράς είναι το συγκεκριμένο άρθρο της συνθήκης, ενισχύεται και η σημασία της συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία θέλει να δημιουργήσει ένα πραγματικό χώρο ελευθερίας δικαιοσύνης και ασφάλειας, ο οποίος θεωρήθηκε από όλους ως μεγάλη καινοτομία στην ε, έναρξη ισχύω της συνθήκη Λισαβόνα. Ευχαριστώ κυρία Ρενάτε Βέμπερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ ε, τις δύο εισηγήτριε, αλλά και τη νομική μας υπηρεσία του Κοινοβουλίου και τον κύριο Περίγιο που νομίζω ότι μας τα παρουσίασε τα θέματα με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια βλέπουμε τις δύο θεωρήσεις, τις δύο σχολές ε, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου εξέφρασε την πιο προηγμένη ας πούμε άποψη και έτσι μπορεί να έχει και αξία για τα θύματα η εντολή αυτή. Εγώ τώρα έχω μερικές ερωτήσεις πάρα πολύ σύντομες νομικής φύσεως διότι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η νομική βάση. Αναφερθήκατε στο άρθρο 3 της συνθήκης. Και αυτή τη διάσταση της πρόληψης της εγκληματικότητας και της καταπολέμησης του εγκλήματος. Αλλά είπατε ότι δεν είναι προληπτικό μέτρο, αλλά είναι μέτρο προστασίας προς ένα πρόσωπο. Πού το βρήκατε αυτό στο άρθρο 3 όμως. Πού το βασίζεται. Και τι σημαίνει αυτό. Η νομική φύση της εντολής προστασίας στις χώρες που εκδίδεται ε, κυριαρχεί και επιβάλλει και σε άλλες χώρες την εκτέλεση. Εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει δυνατότητα ε, άμεση εκτέλεση μια εντολή χωρίς να ε, διέλθουμε ε, από όλε τι διαδικασίε και όλα τα στάδια. Εντάξει, το θύμα παραμένει θύμα σε όλη τη ζωή του. Αλλά είναι σημαντικό να το καταλάβω πώς θα έχει η διαδικασία. Και σε ό,τι αφορά τώρα τον ορισμό του ιονή θύματος, Τι θα πει, δηλαδή εγώ πρέπει να αποδείξω ε, αν κάποιος με απειλεί, ας πούμε δέχομαι απειλές κατά της ζωής για να καταλάβετε ότι είμαι θύμα πρέπει να με σκοτώσουν ή πρέπει να νοσηλευτώ για έξι μήνες για να εκδοθεί τέτοια εντολή, για να καταλάβουν ότι είμαι θύμα. Αυτά ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστώ. Ρομέρο. Ευχαριστώ κύριος Ρωμέβα Ιρουέδα. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε πόσο επίκαιρη ήταν ε, η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, διότι αυτή τη στιγμή μας δίνονται τεράστιες ευκαιρίες να συνεχίσουμε το έργο μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν οικοδομείται μόνο από αυτά τα οποία είναι δυνατά, αλλά και από αυτά τα οποία είναι απαραίτητα. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια ανάγκη και νομίζω ότι ως προς αυτό συμφωνούμε όλοι. Επίσης, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι γνωστό της πάση, πόσο δύσκολη είναι η εκτέλεση μιας απόφασης. Και φυσικά οι διαφορές και η περιπλοκότητα η οποία προκύπτει από την εφαρμογή μιας εντολής σαν αυτή την οποία συζητάμε. Γι' αυτό ακριβώς και χαιρετίζω την έκθεση των δύο συνεισηγητριών, διότι θεωρώ ότι πραγματικά μας δίνουν ένα νέο τρόπο να αναζητήσουμε την ευελιξία η οποία θα μας επιτρέψει να βρούμε μία λύση για τις δυσκολίες που ανακύπτουν. Και νομίζω ότι αυτό το κάνουν κατά τρόπον ώστε να υποχρεούμεθα εμείς ως ε, νομοθέτες ή συνομοθέτες αν θέλετε να αναλάβουμε την ευθύνη να διευκρινίζουμε τα πράγματα εκ των προτέρων και όχι το θύμα να είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να το κάνει. Το θύμα άλλωστε έχει τη μικρότερη υποχρέωση να τηρεί αυτές τις υποχρεώσεις. Θεωρώ ότι το σημαντικό στοιχείο που προκύπτει και από την έκθεση και από την νομική γνωμοδότηση είναι ότι είμαστε σε σωστή άγουσα. Σαφώς υπάρχουν προβλήματα τα οποία χρήσουν επίλυσης ακόμα, αλλά ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και το Συμβούλιο και τις 12 χώρες οι οποίες προχώρησαν το θέμα αυτό και Επίσης, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν κατάλαβα καλά, αντιμετωπίζει με τη δέουσα ευελιξία το θέμα. Θεωρώ ότι ήταν σφάλμα να προσπαθήσουμε να λύσουμε το θέμα αυτό από δικαστική οδό και θα ήταν πραγματικά επονίδει στο μήνυμα να στείλουμε στην κοινή γνώμη ε, ότι προσπαθούμε να λύσουμε το θέμα κατά αυτόν τον τρόπο, διότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το θέμα αυτό. Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλέ εκκρομότητε ακόμα, αλλά θα ήθελα να διευκρινίσω τη θέση τη ομάδα μα. Θέλουμε να προχωρήσουμε προ αυτήν την κατεύθυνση και θα θέλουμε να υιοθετήσουμε το συντομότερο δυνατόν ένα κείμενο το οποίο θα μα επιτρέψει να είμαστε αποτελεσματικοί. Θα ήθελα να ολοκληρώσω με ένα σύντομο συμπέρασμα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να μας πείσει όλους και όλες ότι έχουμε την κατάλληλη νομική βάση για να δράσουμε είναι αυτό το οποίο είπε η νομική υπηρεσία με το οποίο συμφωνώ είναι το άρθρο 3 της συνθήκης. Οι συνθήκες διευκρινίζουν την υποχρέωση των θεσμικών οργάνων να διασφαλίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία με ασφάλεια και ελευθερία. Και αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι το άρθρο το οποίο θα πρέπει να αποτελεί το κίνητρο για τις δράσεις μας. Δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε με άλλα θέματα, τα οποία ναι είναι περίπλοκα και πρέπει να λύσουμε, αλλά δεν είναι τοσιώδες αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ κύριε Ρωμέβα. Η κυρία Κορνίλια Ένστ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχά θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τη νομική υπηρεσία που τόσο νωρίς και εγκαίρως μας ε, διαφώτισε και μας ενημέρωσε για τη νομική αφετηρία και βάση. Και πραγματικά με καθησυχάζει αυτό που ακούω ότι υπάρχει βεβαίως νομική βάση και επαρκής και το άρθρο 3 το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό που είπατε γιατί καταλαβαίνουμε ακριβώ τι σημαίνει χώρο ελευθερία. Να το πω ξεκάθαρα. Όταν κάποιο απειλείται και πάει σε ένα άλλο κράτο μέλος, από το κράτο που έχει εκδοθεί η εντολή προστασίας δεν μπορεί να προστατευτεί, τότε αυτό δεν νοείται ω χώρο ελευθερία. Και έτσι, εκεί θα πρέπει να το βλέπουμε. Ε, η προστασία είναι προτεραιότητα. Η προστασία του απειλουμένου προσώπου θα πρέπει να μας καθοδηγεί στην προσπάθεια αυτή. Γι' αυτό ευχαριστώ και τις δύο εισηγήτριες που μπήκαν πραγματικά σε ε, παρθένο έδαφος και χρειάστηκε και μεγάλη εξερεύνηση ε, και από τις δύο πλευρές και με μεγάλη προσήλωση. Ευχαριστώ πολύ ε, για την προσέγγιση αυτή. Τώρα, κάτι άλλο που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και το θεωρώ σημαντικό. Καταλαβαίνω ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Από τη μια έχουμε διαφορετικά δικαιικά συστήματα και ένωμη τάξη σε κάθε χώρα. Από την άλλη όμως έχουμε ένα μέλημα ε, σε ε, ευρωπαϊκό επίπεδο να γίνει αυτή η προσπάθεια. Παντού ίδια. Και γι' αυτό θα πρέπει να ορίσουμε ξεκάθαρα ποια πρόσωπα είναι αυτά που απειλούνται. Θα πρέπει πολύ συγκεκριμένα να αναγράφονται ε, να κατονομάζονται οι κατηγορίες των προσώπων για να μπορεί να έχει και εφαρμογή αυτή η εντολή. Και επίσης ποιες είναι οι αξιόπινες πράξεις ή ποιες είναι οι απειλές που καλύπτονται. Ε, και η ψυχική παρενόχληση και η ηθική παρενόχληση ανήκει εδώ και το stalking ακόμα. Όταν κάποιος καταδιώκει ένα θύμα και βεβαίως και μια κατηγορία μαρτύρων, προστασία των μαρτύρων που είναι μια κατηγορία πάρα πολύ ε, ιδιαίτερη που απειλείται πάρα πολύ. Αυτά είναι κάποια σημεία που χρειάζονται περισσότερη πρόσοχη. Επίσης θα πρέπει να δοθεί ε, προστασία ανεξάρτητα ε, από την αρμοδιότητα. Είναι αυτά τα ζητήματα ποινικά, αστικά ή ακόμα και διοικητικά. Διότι σε τελική ανάλυση μπορεί να υπάρχει διαφορά νομική, αλλά στην ουσία όταν κάποιος απειλείται, απειλείται, δεν έχει σχέση με το τι δικαστήριο είναι αυτό. Δεν συμφωνώ να έχουμε διαφορετικές οδηγίες, ε, άλλοι για το ποινικό σκέλος, άλλοι για το αστικό σκέλος, όχι. Είναι δύσκολο για μένα να το διαχωρίσουμε, γιατί αλλοιώνει και τα δικαιώματα ε, των ε, θυμάτων και τα κατακαιρματίζει. Και δεν μου αρέσει αυτό. Και ένα άλλο θέμα που θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό, εκτός από τροπολογίες βεβαίως που θα κάνουμε και εμείς ως ομάδα, θέλω να τονίσω το εξής. Τα πρόσωπα που απειλούνται θα πρέπει να ενημερώνονται για όλα τα μέτρα προστασίας τους στα πλαίσια της εντολής, αλλά δεν θέλουμε Ε, να ε, διαδίδονται αυτές οι πληροφορίες, δηλαδή να ενημερώνονται οι ενδιαφερομένοι, αλλά όχι και ο περίγυρός τους, ας πούμε, και τα κοντινά τους πρόσωπα. Θα κάνουμε τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή. Ε, λοιπόν, ένα τελευταίο. Η εντολή προστασίας λέει που θα πρέπει να ισχύει μόνο εφόσον είναι κάποιος αποδεδειγμένα θύμα. Μα αυτό τι προστασία είναι και τι εντολή προστασία. Είναι πολύ κοντόφθαλμο αυτό. Θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι, πολύ να προσέξουμε πώς θα είναι το πεδίο εφαρμογής αυτής της εντολής. Και συμφωνούμε με το Συμβούλιο. Πρέπει να βελτιωθεί αυτό. Ελπίζω να καταλήξουμε σε μια κοινή λύση. Danke. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να εφαρμοστεί η Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας μόνο όταν έχει ήδη χορηγηθεί η Εθνική Εντολή Προστασίας. Και δεύτερον, το δικαστήριο στη δεύτερη-τρίτη χώρα ε, δεν μπορεί παρά να χορηγήσει το ΕΠΟ εφόσον έχει εκδοθεί η Εθνική Εντολή στο πρώτο κράτος μέλος. Άρα αναρωτιόμαστε ποιο είναι το πεδίο του ορισμού της εντολής. Ε, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό διότι είναι εφαρμοστέα διαφορετικά ένομα συστήματα στο πρώτο ή στο δεύτερο κράτος μέλος. Επίσης, ε, απεδείχθη ότι αυτός ε, που ισχυριζόμαστε ότι συνιστά κίνδυνο θα πρέπει να καλυφθεί από την εφαρμογή του ΕΠΟ. ο δράστης αυτός ε, που συνιστά κίνδυνο ε, με την εντολή προστασίας επειδή ενημερώνεται για την έκδοση ε, της εντολής προστασίας θα γνωρίζει που πήγε το ιονή θύμα. Και το, ο άλλος επιπρόσθετος κίνδυνος ε, είναι ότι ο δραστής ή αυτός ε, που απειλεί μπορεί να ισχυριστεί ότι ε, βρέθηκε τυχαία στο ίδιο κράτος με το Ιωνί θύμα. Βέβαια είναι γελίο αυτό. αν σκεφτεί κανείς ότι προέρχεται ο δράστης και το θύμα από την ίδια πόλη, από το ίδιο κράτος. Άρα, Αντί να έχουμε νέα ευρωπαϊκή εντολή, καλύτερα θα ήταν όταν ε, υπάρχει παραβίαση της αρχικής εντολής να ε, ε, εκδοθεί εντολή για το δράση να επιστρέψει στο πρώτο κράτος μέλος. Οπότε το δικαστήριο εκεί να αποφασίσει αν πρέπει να τροποποιήσει το πεδίο της αρχικής εντολής. Βέβαια καταλαβαίνω ότι αυτό είναι στα πρόβλημα, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει και μία τάση να χρησιμοποιούμε ε, πραγματικά ε, προβλήματα για να επεκτείνουμε τις δικαστικές αρμοδιότητες της Ένωσης ε, ανά την επικράτειά της. Ευχαριστούμε κύριε Μαλικόβεϊ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαι η σκιώδης εισηγήτρια της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για αυτό το σχέδιο και εν συντομία θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία ζητήματα. Πρώτον, τροπολογία 15 όπου προβλέπεται ότι κατά την εφαρμογή αυτής της οδηγίας θα πρέπει να θεσπίσουν διαδικασίες στα κράτη-μέλη, ούτως ώστε ο προστατευόμενος και αυτός που συνιστά κίνδυνο να καταθέσουν μαρτυρία στο νέο κράτος, έτσι, στο κράτος εκτέλεσης. Αυτό αντιβαίνει στο πεδίο και στο στόχο της οδηγίας, ε, δηλαδή την εσπεσμένη προστασία του θύματος. Επίσης ε, δεν έχει και πάρα πολύ νόημα γιατί ο προστατευόμενος είναι αυτός που ήδη έχει ε, υποβάλει έτοιμα για την προστασία. Δεν χρειάζεται εκ νέου ακροασή Στην τροπολογία 13 προβλέπεται επίσης υποχρέωση Ενημέρωση των ε, δύο μερών των διαδίκων για το μέτρο. Οπότε θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά αυτή τη διαδικασία. Δεύτερον, τροπολογία 10. Εκεί αναφερόμαστε ε, στη δυνατότητα που έχει το κράτος εκτέλεσης ε, να εγκρίνει μέτρα, και τώρα παραθέτω, ενιολογικά και νομικά ανεξάρτητα από το αρχικό μέτρο προστασίας ε, του κράτους έκδοσης της εντολής. Ε, και αυτό είναι επικίνδυνο ενδεχομένως ε, γιατί προσθέτει έτσι μία έννοια ευθερετότητα στην απόφαση και αν ε, θεσπιστεί ε, εντελώ ε, νέο μέτρο θα πρέπει να κινηθεί άλλη διαδικασία κατά αυτού που συνιστά κίνδυνο. Οπότε νομίζω είναι αιτιολογημένη η ανησυχία στον τομέα αυτό. Τρίτον, Έχουμε ακούσει διεστάμενες απόψεις και γι' αυτό αναφέρομαι σε αυτό. Το potential victims, οι θύματα, αυτή την ορολογία που χρησιμοποιούμε. όρο. Υπάρχει ορισμός για το θύμα. Ε, υπάρχει ορισμός όπου νομικός πώς θεωρείται κάποιο θύμα. Τώρα, αυτό το potential, ο χαρακτηρισμός ή possible victim, πιθανό θύμα, δεν ε, ε, συνάδουν με την νομή, τη διατύπωση της νομικής πράξης. Δηλαδή, όταν προστατεύεται κάποιος με την εντολή, τότε γίνεται θύμα. Άρα, ε, τι, ενδυνάμει θύματα είναι όλοι που βρίσκονται κάπου, οπουδήποτε και που ενδεχομένως μπορούν να υποστούν επίθεση. Δεν είναι νομική έννοια αυτό το ενδυνάμει θύμα. Ευχαριστούμε η Σίλβια Κώστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως ε, σκιώδης εισηγήτρια της Επιτροπής Γυναικών θα ήθελα να ευχαριστήσω τις δύο εισηγήτριες οι οποίες έκανε πολύ καλή δουλειά από κοινού, ε, γεγονός που αποστέλει ένα στεναρό μήνυμα από πλευρά συνεργασίας των δύο επιτροπών και ξεκινά και τις κοινέ αυτές ε, συνεδριάσεις. Να ευχαριστήσω επίσης την νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία μας είπε σαφώς ποιες είναι οι πιο θαραλές ερμηνείες που μπορούμε να δώσουμε ε, και νομίζω ότι περιέχονται και στις τροπολογίες των δύο συνεισηγητριών, όχι μόνο ως προς την νομιμότητα της νομικής βάσης, αλλά και ω προ το γεγονό ότι η διαδικασία αυτή είναι πιο ευρεία από ό,τι προβλέπεται στο αρχικό κείμενο. Η παράγραφο ε, Δ του άρθρου 82, αλλά και η παράγραφο άρθρα, αλλά και η πιο κατάλληλη ερμηνεία του άρθρου 3 τη συνθήκη τη ε, Λισαβόνα. Νομίζω ότι αυτό θέτει εκ νέου το θέμα στη βάση της αμοιβαιότητας ε, των αποφάσεων που εκδίδονται από ένα κράτος μέλος και το σεβασμό τους από άλλο κράτος μέλος και επίσης συζητά το θέμα του δικαιώματος του ανθρώπου ως πολίτης, ως ε, πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τη χάνει προστασίας από δυνητικές εγκληματικές ενέργειες και νομίζω ότι αυτό ενισχύει πολύ περισσότερο ε, την απόπειρα αυτή που κάνουμε. Επίσης, εγώ είμαι σκιώδη εισηγήτρια για την Επιτροπή Γυναικών και θα πρέπει να διευκρινίσω ότι εδώ μιλάμε για εντολέ προστασία που δεν αφορούν μόνο τι γυναίκε, Επειδή παρά το γεγονό ότι γνωρίζουμε ότι οι γυναίκε είναι αυτέ οι οποίε στατιστικά ε, είναι τα περισσότερα θύματα, μιλάμε και για του ανηλίκου και εδώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τις συνεισηγήτριες διότι επισήμαναν πόσο σημαντική είναι η μέρημνα για τους αλληλίκους και τους ε, ε, δαιμόνες τους ε, όταν υπάρχει εντολή προστασίας, ε, το οικογενειακό περιβάλλον το οποίο λαμβάνεται υπόψη και επίσης έχουμε και άλλα ιονή θύματα. Αναφέρθηκε για παράδειγμα το θέμα των μαρτύρων ή κάποιων άλλων που είναι δυνητικά θύματα και χαίρομαι ιδιαίτερα που το κείμενο αναφέρεται σε πρόσωπα και δεν κάνει μια καταγοριοποίηση η οποία κατά την άποψή μου δεν θα είχε καμία χρησιμότητα αυτή τη στιγμή κάτι επιπλέον, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσω και πάλι τις συνεισηγήτριες, ε, το γεγονός ότι έλαβαν υπόψη όλες τις παρατηρήσεις μας για την πραγματική πρόσβαση για θύματα τα οποία ήδη έχουν μία εντολή προστασίας και είναι σημαντικό να γνωρίζουν ε, πόσο αποτελεσματική είναι αυτή η εντολή και ε, να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες. Αυτός ο ευρωπαϊκός αριθμός που προτείνεται, στον οποίο αναφερόμαστε πολύ συχνά και είναι πολύ ενδιαφέρον να μπορέσουμε να έχουμε έναν ε, αριθμό στον οποίο κάποιος μπορεί να καλέσει και να λάβει πληροφορίες ε, για το κατά πόσον μπορεί να εφαρμοστεί μια εντολή προστασίας. Και το θύμα λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα έχει δικαίωμα σε προστασία εάν μετικήσει σε άλλη χώρα μέρα. Αλλιώ είναι πάρα πολύ δύσκολο να γνωρίζει ότι έχει αυτό το δικαίωμα. Τρίτον, είναι πολύ σημαντικό το γεγονό ότι θα πρέπει να είναι δωρεάν η πρόσβαση σε αυτό το μέσο και επίση θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία υποχρέωση ενημέρωση και για το θύμα αλλά και για το θήτη. Να σας πω για παράδειγμα ότι στην χώρα μου, στην Ιταλία, όπου εισήχθη η εντολή προστασίας και για θέματα stalking και μόνο το γεγονός ότι υπάρχει ενημέρωση προς το θήτη και το γεγονός ότι γνωρίζει ότι τον προσέχουμε και προσέχουμε τις συμπεριφερές του άλλαξε πάρα πολύ το τοπίο και ελπίζω ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει τη θέση της επί του θέματος, διότι έχει βάλει στο επίκεντρο το θέμα της προστασίας του θύματος ε, και όχι μόνο την ε, αναγνώριση μεταξύ διαφορετικών δικαστικών, ποινικών και αστικών συστημάτων. Ευχαριστώ. Έχουμε ένα ακόμα αγορητή, η κυρία Μαρίνα Γιανακουδέκης αλλά δυστυχώς έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ με την πρωινή ημερήσια διάταξη, γι' αυτό σας παρακαλώ να είστε λακωνικοί, διότι έχουμε κι άλλη κοινή συνεδρίαση. Σας παρακαλώ λοιπόν να είστε σύντομοι. Θα είμαι πολύ γρήγορη, εξαιρετική ιδέα, μπορούμε να συνεργαστούμε. Ναι. για αυτή την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Υπάρχουν πολλοί προβληματικοί τομείς όμως. Ε, θα ήθελα να διευρυνθεί για να ε, καλύπτει όχι μόνο την προστασία αλλά την εμπορία ανθρώπων, τη βία κατά των αντρών, ε, την κακοποίηση παιδιών. Λοιπόν, για να λειτουργήσει το σύστημα πρέπει να έχουμε ισχυρή νομοθεσία, κρατέα νομοθεσία και από ό,τι άκουσα δεν είναι αρκετά ισχυρή η νομική βάση σήμερα και η συναδέλφο, ο συναδέλφός μου είπε ότι δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για την νομική βάση, γιατί ε, περί τίνος πρόκειται για την προστασία του θύματος. Ε, το θύμα είναι κάποιος που ορισμού δεν έχει εμπιστοσύνη στο σύστημα, νιώθει ανασφάλεια. Δεν θα νιώσουν καλύτερα επειδή έχουμε την νομοθεσία. Δεν βοηθάει αυτό το θύμα. Επίση, το να θεσπίσουμε αυτή την νομοθεσία που δεν θα λειτουργήσει σε όλε τι ε, χώρε, ε, τελικά θα δημιουργηθούν φρούδε ελπίδε για τα θύματα. Ε, και άρα το θύμα μπορεί να διατρέξει μεγαλύτερο κίνδυνο, γιατί θα πάει κάπου αλλού και θα νομίζει ότι το προστατεύει το άλλο κράτος μέλος, ενώ δεν ισχύει αυτό. Λοιπόν, για να γίνουν όλα σωστά πρέπει να δαπανίσουμε περισσότερο χρόνο στην εξέταση των ζήτημάτων. Νομίζω ότι βιαστήκαμε υπερβολικά. Πρόεδρος, ευχαριστούμε για, όλα αυτά, για όλες αυτές τις παρατηρήσεις και για την προσπάθεια που έκανε η νομική υπηρεσία. Τώρα θα ακούσουμε τον 6ο ε, Πρίλο και πάλι για να απαντήσει ε, σε κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα. Παρακαλώ να είστε και εσείς σύντομος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο, μάλιστα. Σύντομα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα όσα είπατε. Ε, για τη νομική μας υπηρεσία και τη γνωμοδότησή της. Δεν ξέρω, πριν βγω από την αίθουσα, μήπως χρειαστεί ο πρόεδρος να εκδώσει εντολή προστασίας μου. Αλλά ας το κινδυνεύσω και αυτό, τι να κάνω. Η πρώτη ερώτηση ε, που έθεσε κάποιες αφιβολίες είναι η ερώτηση του κυρίου Κίρκοπ για τη νομική βάση. Και είπε ότι υπάρχουν πολλές επιπλοκές στην οδηγία αυτή και διερωτάται και εκείνος ε, το τι εστί ιονή θύμα. Δεν ε, θα λύσει κανείς τα προβλήματα ε, προσθέτοντας και νέες επιπλοκές ή νέες δυσκολίες. Είναι αρκετά δύσκολα από τη φύση τους και είπαμε ότι είναι καινοτόμα αυτή η προσπάθεια. θα γίνουν και τροπολογίες. Λοιπόν, επαναλαμβάνω για το, την έννοια του Ιωνί θύματος. Η εντολή προστασίας βασίζεται σε μια εθνική δικαστική απόφαση, σε μια εθνική αρχή λοιπόν. Η αρχή, η εθνική ε, που αξιολογεί το αν ε, κατά πόσο χρειάζεται να εκδοθεί μια εντολή προστασίας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει αυτή η εθνική εντολή, μπορεί να προσθεθεί και μια ευρωπαϊκή ε, κατ' επέκταση, ακριβώς για να επιτρέπει αυτή τη διεύρυνση της προστασίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκρισμπέκ που είπε ότι είναι πολύ καλή ιδέα. Εγώ δεν διεκδικώ την πατρότητα. Η ίδια η οδηγία το ορίζει αυτό. Ότι η εντολή προστασίας εκδίδεται με στόχο τη ε, συνέχιση της ε, προστασίας και της ασφάλειας του προστατευομένου προσώπου. Εγώ απλώς και μόνο εφαρμόζω ε, αυτή την ιδέα στην πρότασή μας. Η κυρία Βέμπερ μας ρώτησε τι γίνεται ακριβώς με το άρθρο 3. Αν θα πρέπει να δανειστούμε το τμήμα που αναφέρεται στην πρόληψη ή το τμήμα που αναφέρεται στην προστασία. Εδώ, στο ποινικό δίκαιο, πρόκειται για προστασία, αλλά η άλλη όψη του νομίσματος είναι και η πρόληψη. Γιατί μιλούμε για επιθετικές ε, πράξεις, ε, ενδεχομένω και εγκληματικές. Εδώ όμως δεν είναι ε, αυτό το ζητούμενο. Είναι η προστασία προτεραιότητα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το άρθρο 84 της συνθήκης προβλέπει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε συναπόφαση να ορίσουν μέτρα που θα ενθαρρύνουν ή θα υποστηρίζουν τη τράση των κρατών μελών στον τομέα της πρόληψης του εγκλήματος. Πρόληψη εγκλήματος εδώ εννοείται διασυνοριακό, έτσι όπως είναι το οργανωμένο έγκλημα, οι μαφίες κτλ. Από τη φύση του λοιπόν και μόνο αυτό το έγκλημα είναι διασυνοριακό. Ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση για τα θύματα είναι εδώ οικογενειακή βία. Δεν έχει καμία διασυνοριακή χρειά η φύση του εγκλήματος. Αντίθετα, το, το πρόσωπο είναι εκείνο που χρήζει προστασίας και όταν μετακινείται. Όταν κάποιο λοιπόν εκτίθεται σε μια απειλή επίθεση ενδοοικογενειακή στην Ιταλία, το ίδιο πρόσωπο θα πρέπει να προστατεύεται και αλλού. Αυτή τη στιγμή ε, μεταβεί σε ένα άλλο κράτος μέλος, όπου παραμένει ο κίνδυνος. Έτσι, γι' αυτό ακριβώ το λόγο θεωρούμε, θα δούμε όμω, γιατί δεν έχουμε και το μονοπόλιο, δεν κατέχουμε εμεί την αλήθεια, ε, να δούμε λοιπόν πώς αυτή η εντολή θα ε, εγγραφεί σε μια νέα ελευθερία που είναι η ελευθερία να κυκλοφορεί κανείς σε ένα χώρο ασφάλειας, δικαιοσύνης και ελευθερίας. Και αυτή είναι μια επανάσταση της ε, συνθήκης Λισαβόνας που καθιστά πλέον κοινοτική όλη τη διάσταση του τρίτου πυλώνα του παλαιότερου. Τελειώνω με την εξής παρατήρηση. Είπε κάτι η κυρία Κώστα, ενδιαφέρον, από πλευράς αξιολόγηση της εντολής αυτής. Είπε η κυρία Κώστα ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι γυναίκες και οι ανήλικοι βεβαίως, αλλά και οι μάρτυρες να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το πρόβλημα. Δυστυχώς, η εντολή, δυστυχώς, Ευτυχώς θα έλεγα. Ευτυχώς. Η εντολή προστασία ακριβώς δεν αφορά την προστασία των μαρτύρων. Σαφέστατα ορίζεται αυτό. Για τον εξής απλούστατο λόγο. Οι μάρτυρες θα πρέπει να προστατεύονται βάσει της μαρτυρίας τους, της μαρτυρικής τους κατάθεσης. Ε, εδώ η προστασία αφορά ένα πρόσωπο που απειλείται δεν, είναι, δεν έχει να κάνει με μια μαρτυρική κατάθεση. Από το γεγονός ας πούμε ότι είναι ένα πρόσωπο γυναίκα απειλείται και μόνο ε, από αυτό όχι επειδή κατέθεσε κάτι ή έδωσε μια πληροφορία ή είχε μια συμπεριφορά απέναντι στη δικαιοσύνη. Είναι από, από την ύπαρξή της και μόνο ε, που απειλείται και καλεί την προστασία σε κάποιες ε, δεδομένες συνθήκες. Και ένα τελευταίο τώρα για το θέμα της αναγνώρισης που έλεγε η κυρία Βέμπερ. και που αποκλείσαμε ως αναγνώριση αμοιβαία δικαστικών αποφάσεων. Στο άρθρο 9 η οδηγία ομιλεί για αναγνώριση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας και αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, οι δικαστές του κράτους εκτέλεσης της απόφασης του άλλου ε, από εκείνο που έχει εκδοθεί καλούνται να εξετάσουν ε, αυτό το στοιχείο από την ευρωπαϊκή πλευρά και όχι από την αμοιβαία διμερή αναγνώριση. Δεν υπάρχει πλέον η διακυβερνητική διάσταση, αφού είναι κοινοτική πλέον. Το άρθρο 9 λοιπόν θα πρέπει βεβαίως να εξακριβώνεται βάσει το άρθρο 9 αν ε, προκύπτει αυτή η περίπτωση και βρίσκει εφαρμογή και είναι ευρωπαϊκή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστούμε κύριε Περίλο. Να σας υπενθυμίσουμε ότι η προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών είναι 9 Ιουνίου 12 το μεσημέρι. Να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη τα οποία συνεισέφεραν στο θέμα αυτό. Μας πιέζει ο χρόνος να περάσουμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Το σημείο υπαριθμών 14. Θα θυμάστε ότι το 13 ακυρώθηκε. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε στη θέσπιξη ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαγύγιο και το δικαστικό χωρισμό. Το περιβόητο Ρώμη 3. And jury committees work together είναι κοινή συνεργασία της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και της Επιτροπής Γιούρη. Θα θυμάστε ότι τον Οκτώβριο του 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε στη διαδικασία της ε, ε, διαβούλευσης στην γνωμοδότησή του ε, διαδικασία στην οποία εγκρίθηκε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πλέον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει στη διαδικασία διαβούλευσης για μια απόφαση που εγκρίνει την ενισχυμένη συνεργασία για το θέμα αυτό. Η ενισχυμένη συνεργασία προκύπτει βάσει της συγκεκριμένης διαδικασίας της συνθήκης επειδή δεν υπήρχε συνένεση στο Συμβούλιο. Θα ακούσουμε τώρα την έκθεση της κυρίας Γκέπχαρτ. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα μπω σήμερα στην ουσία των θεμάτων γιατί στις 10 του μηνός ε, θα τα συζητήσουμε ε, με μεγαλύτερη ε, χρονική άνεση. Θα ήθελα να σας εξηγήσω λίγο ξανά τη διαδικασία για να γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι περί τίνος πρόκειται. Όντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έτος 2006 έκανε μια πρόταση νομοθετικού περιεχομένου βάσει των συνθηκών τότε της Νίκαιας, βέβαια και της Συνδίκης της Λισαβόνας, ε, στον τομέα του οικογενειακού δικαίου έχουμε αμοιβέ αναγνωρίσεις σε αυτούς ε, τους τομείς και προβλέπεται ομοφωνία στο Συμβούλιο. Απεδείχθη όμως ότι σε αυτά τα θέματα αμοιβαία αναγνώρισης ε, χωρισμών και διαζυγίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια τέτοια ομοφωνία δεν προκύπτει. Είναι, είναι αδύνατο να επιτευχθεί. Γι' αυτό τον Ιούνιο του 2008 σε συνεδρίασή του το Συμβούλιο δήλωσε επίσημα ότι επειδή δεν μπορούμε να πετύχουμε ομοφωνία θα πρέπει να ε, ανασταλεί η διαδικασία. 16 εκατομμύρια ε, ε, ε μικτούς γάμους έχουμε από δύο εθνικότητες συν ε, γάμους ε, ε, πολιτών που ζουν σε μια χώρα διαφορετική από τη δική τους και εργάζονται και χωρισμοί και τα Και δεν είναι πάντα γνωστό ποιος δικαστής είναι αρμόδιος, ποιο δίκαιο εφαρμόζεται Και υπάρχουν ε, ε, ζευγάρια που θέλουν να χωρίσουν αλλά δεν βρίσκουν δικαστή γιατί δεν ξέρουν τι ισχύει και ποιος θα αποφασίσει. Στην περασμένη λοιπόν η θητεία και σε συνεννόηση με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ε, το είχαμε συζητήσει με τον τότε Επίτροπο κύριο Μπαρό. Μήπως χρειάζεται άραγε ενισχυμένη συνεργασία των κρατών μελών έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα για τους πολίτες όσο γίνεται ε, περισσότερο. Γιατί δεν μπορούμε να το αναβάλουμε αυτό στο δινεκές και με τη συνθήκη της Λισαβόνας γνωρίζουμε ότι την επόμενη πενταετία και πάλι δεν πρόκειται να δοθεί λύση σε αυτά τα θέματα. Ε, σύμφωνα λοιπόν με τη συνθήκη της Λισαβόνας, εννέα κράτη θα πρέπει να κάνουν ε, μια τέτοια αίτηση. Όντως έγινε, ζητήθηκε αυτό από εννέα κράτη-μέλη. Γαλλία, ε, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Αυστρία, Ισπανία, Ιταλία, Σλοβενία και Λουξεμβούργο. Ήταν οι εννέα χώρες που υπέβαλαν αυτό το αίτημα. Ακριβώς εννέα. Στο μεταξύ προσθέθηκαν το Βέλγιο, η Λιθουανία και η Γερμανία. Είπαν ότι θέλω να συμφωνήσουν. Η Ελλάδα απεσύρθη, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θα ρωτήσω και θα μάθω και θα σα πω γιατί ε, το ξανασκέφτονται. Είχα και ίδια επαφή με την νομική επιτροπή. Ο κύριος Σβίφκα πρέπει να σας πω είναι πάρα πολύ επικοδομητικός και πρόθυμος για συνεργασία και συζητήσαμε πώς θέλουμε να προχωρήσουμε. Στις 3 και 4 Ιουνίου συνεδριάζει το Συμβούλιο, το οποίο ε, θα ήθελε να αποφασίσει αυτή την ενισχυμένη συνεργασία και χρειάζεται απόφαση της νομικής επιτροπής προηγουμένως. και ελπίζω να συμφωνείτε μαζί μου, είπα ότι δεν ε, είναι ανάγκη να γνωμοθετήσουμε γι' αυτό και μόνο το σημείο της νομικής βάσης, είναι μόνο για τη νομική βάση. Θεώρησα λοιπόν ότι συμφωνούμε ε, να ψηφίσει σήμερα η Επιτροπή μας, η ε, ΛΥΜΠΕ, για να αρχίσει η διαδικασία και να μπορέσουμε επιτέλους να περάσουμε στην ουσία του θέματος. Πάντα σε συνεννόηση μαζί μου Η ενισχυμένη συνεργασία λοιπόν όχι μεταξύ των επιτροπών αλλά ε, για τη διαδικασία αλλά για την ουσία εν πάση Λοιπόν, σήμερα το πρωί στις 10 η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων συνεδρίασε και ψήφισε ε, για την νομική βάση και ομόφωνα συμφώνησε για την ενισχυμένη συνεργασία. Και καλό είναι αυτό, γιατί θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την υπόθεση, να τελειώνουμε και να βρούμε λύσεις. Δεν θέλω να μπω στην ουσία σήμερα, επαναλαμβάνω, ε, θα το κάνουμε αργότερα. Εν ευθέτω χρόνο. Την άλλη εβδομάδα ή την παράλληλη θα συναντήσω τον κύριο Τσβίφκα που είναι ο εισηγητής σας είπα επί της ουσίας στην Νομική Επιτροπή. Αν θέλετε και μετά να τα πούμε με τους κοιόδης εισηγητές της Επιτροπής μας εδώ, Λίμπε, για να σας ενημερώσω αμέσως και μετά στις 10 Ιουνίου μπορούμε με βάση όλα αυτά να μπούμε στην ουσία του θέματος. Μέχρι πού θέλουμε να φτάσουμε. Υπάρχουν ήδη μερικά θέματα προς συζήτηση. Ερχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής μιλούσε για την επιλογή του δικαστή και του δικαίου. Ποιο δίκαιο βρίσκει εφαρμογή ποια χώρας. Το περιόρισε λίγο το Συμβούλιο και θα πρέπει να το συζητήσουμε, να δούμε αν συμφωνούμε με αυτή την υπόθεση, αυτό τον περιορισμό ή θέλουμε κάτι άλλο. Αλλά όπως σας είπα, ήδη αρκετές φορές θα τα πούμε αυτά στις 10 Ιουνίου. Πού θέλουμε να πάμε, μέχρι πού θέλουμε να πάμε κτλ. να δούμε τι θέλει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς τα που θα κινηθούμε. Ελπίζω να προχωρήσουμε. Άτυπα άκουσα στο μεταξύ στο ράδιο Αρβίλα ότι αν αποφασίσει επίσημα στις 3 και 4 ε, Ιουνίου το Συμβούλιο Ενισχυμένη Συνεργασία θα ήταν αυτό πρώτη φορά που θα συμβεί στο ευρωπαϊκό δίκαιο και μετά άλλα τρία κράτη θέλουν να προσθεθούν έτσι κι αλλιώς είναι ανοιχτή η διαδικασία, ανά πάσα στιγμή μπορεί ο καθένας να ε, συνεργαστεί σε αυτή την ενισχυμένη συνεργασία. Και χώρες που δεν είναι αυτή τη στιγμή να ενταχθούν στο σύστημα. Για να μην έχουμε δίκαιο πρώτης κατηγορίας και δεύτερης κατηγορίας να μπουν όλες οι χώρες που το επιθυμούν. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπουν και 27. Αυτό ελέγχεται. Ούτε είναι του παρόντος. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκέπχαρτ που μας παρουσιάσατε την κατάσταση για αυτή την ενισχυμένη συνεργασία. Εξ όσο γνωρίζω, ούτε η Προεδρία ούτε η Κομισιόν θέλουν να λάβουν τον λόγο. Να μην χρειάζεται κιόλα. Η κυρία Αντζελίλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκέπχαρτ για την παρουσίαση αυτή και ήθελα να προσθέσω και κάποια στοιχεία που μας δίνουν μια εικόνα του πόσο σημαντική είναι αυτή η νομοθεσία. Τα επίσημα στοιχεία μας λένε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε περίπου 300.000 διεθνείς ε, γάμους ετησίως. Μιλάμε για γάμους, δηλαδή για ενώσεις οι οποίες αναγνωρίζονται νομικώς. Υπάρχουν και άλλες μορφές βέβαια ένωσης, γάμου. Πρόκειται λοιπόν για ένα θέμα το οποίο στην ε, εφαρμοστέα νομοθεσία διαζυγίων και ε, δικαστικών χωρισμών αφορά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό κρατώ, ε, πολιτών. Καλώς λοιπόν τα εννέα κράτη-μέλη ζήτησαν ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα αυτό. Πρόκειται για την πρώτη φορά στην οποία θα υπάρχει αυτή η διαδικασία, διότι το θέμα είναι κατεπήγον. Ο Ευρωπαίος νομοθέτης έχει καθυστερήσει. Τον έχουν προλάβει τα γεγονότα. Αυτό λοιπόν το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι την ύφη για αυτό το νομοθετικό κενό την πληρώνουν φυσικά ε, τα ευάλωτα μέρη. Πολύ συχνά είναι οι γυναίκες αυτές οι οποίες ε, πλήττονται και πολύ συχνά φυσικά είναι και οι ανήλικοι. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά η κυρία Γκέπχαρ το θέμα, διότι πέρσι ε, ήταν ε, η εισηγήτρια για την ε, νομοθεσία ε, και το τι ακριβώς γίνεται με τους μικτούς αυτούς γάμους. Αυτή τη φορά βλέπουμε ότι κάθε χρόνο έχουμε χιλιάδες παιδιά τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαμάχης μεταξύ των δύο ε, πρώην συζύγων και ορισμένες φορές έχουμε και απαγωγή. Ο ένας εκ των δύο γονιών δεν έχει πλέον ε, κανένα στοιχείο για το πού βρίσκεται το παιδί του διότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχουν επαρκή μέσα για να διαχειριστούμε αυτή την κατεπίδουσα κατάσταση. Ολοκληρώνοντας να πω ότι μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα η απόπειρα να αυξηθεί ευελιξία στον τομέα αυτό και να ενθαρρύνουμε όπου υπάρχει δυνατότητα ε, τις ε, φιλικές συνενετικές λύσεις οι οποίες μας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσουμε τη διαμεσολάβηση ως ε, προνομιακό μέσο. Αλλιώς έχουμε μια σειρά από φαινόμενα όπως για παράδειγμα στην δικαστική διαμάχη όταν ε, κάποιος εκ των δύο συζύγων θέλει να χωρίσει για να έχει όσο το δυνατόν ε, μεγαλύτερο πλεονέκτημα προσπαθεί ουσιαστικά να ε, είναι ο πρώτος ο οποίος θα προσφύγει στο δικαστήριο ώστε να έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να έχει περισσότερα δικαιώματα πάνω στα παιδιά του. Πρόκειται για μια συμπεριφορά την οποία θα πρέπει να αποθαρρύνουμε με την ομοθεσία μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Ινετβέλτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που έχουμε ξανά εισηγήτρια την κυρία Γκέπχαρτ. Είχαμε συνεργαστεί πολύ καλά για το θέμα αυτό στην προηγούμενη θητεία. Θα ήθελα να υποστηρίξω την πρότασή της, αλλά πρέπει να σας πω με βαριά καρδιά. Γιατί όλοι θα θέλαμε φυσικά ευρωπαϊκή λύση, πανευρωπαϊκή λύση. Τώρα αυτό είναι οπισθοδρόμηση. Και ένα ήταν το κράτος μέλος Μπορεί να είχε ευγενεί στόχους, αλλά τορπίλησε την όλη υπόθεση. Στο μεταξύ έχω δει αρκετές ε, τέτοιες υποθέσεις, γυναίκες όπως είπατε, που έχουν πέσει θύματα σε αυτή την υπόθεση. Και το διαζύγιο ε, έγινε χωρισμός με πολύ αρνητικό τρόπο. Είμαι πάρα πολύ θλιμμένη λοιπόν για αυτή την κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι είναι ένα βήμα προς μια πλήρη πανευρωπαϊκή κάλυψη και λύση, γιατί πιστεύω ότι με το γεγονός να αρνηθούμε τότε την ε, ρύθμιση δεν μειώθηκαν τα διαζύγια. Αλλά τα διαζύγια παρέμειναν με κακές συνθήκες να εκδίδονται. Έτσι, θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός. Έχω μερικές ερωτήσεις. Εγώ δεν είμαι συνταγματολόγος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πόσο επηρεάζει εδώ ακόμα. Γιατί έχω και άλλη ερώτηση. Ε, είπατε ότι το Συμβούλιο περιόρισε ακόμα περισσότερο το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία και εμεί θέλουμε να το διευρύνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε ή απλώ το προτείνουμε έτσι γενικά. Και κάτι άλλο που είμαι περίεργη γι' αυτό αν εγκριθεί αυτή η ενισχυμένη συνεργασία, υπάρχουν άλλα τρία κράτη-μέλη που είναι πρόθυμα να προσχωρήσουν. Και είχα την περιέργεια να μάθω ποια είναι αυτά τα τρία. Ελπίζω το δικό μου κράτος να δείξει αυτή τη φρόνηση και τη σύνεση να προσθεθεί. Και θα έχουμε και σε δύο εβδομάδες νέα κυβέρνηση, να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ανήκει και το δικό μου κόμμα σε αυτή φυσικά. Members Ευχαριστώ. Δεν θα ήθελε κανένας άλλος το λόγο από ό,τι βλέπω. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε γιατί ήσασταν σύντομοι και μας βοηθήσατε να προλάβουμε, να τελειώσουμε την ημερήσια διάταξη. Ευχαριστούμε κυρία Γκέπχαρτ για την ε, παρουσίαση. και θα ε, περιμένουμε νέα σας. Πολύ σύντομα. Δεν θέλω να σας πάω χρόνο. Για αυτά που είπε η κυρία Αντζελίλη και η κυρία Νετβέλτ, η Σόφη, αυτό που πρέπει να αποφύγουμε είναι αυτό το shopping που υπάρχει σήμερα, που μπορεί ο καθένας να επιλέγει πού θα πάει και τι θα κάνει, και αυτό είναι εις βάρος των γυναικών τελικά. Και ακριβώ ότι δεν υπάρχει και αμοιβαία αναγνώριση των διαζυγίων των δικαστικών χωρισμών. Είναι πολύ σημαντικό να ρυθμιστεί αυτό. Για αυτά που είπε η Σοφή, ποιε είναι οι τρει χώρε, δεν μπορώ να σα αποκαλύψω σήμερα ακόμα. Καμιά φορά έχουμε εμπιστευτικέ πληροφορίε, αλλά επιθυμώ να το κοινοποιήσουν οι ίδιε οι χώρε. Δεν θέλω να το πω εγώ. Και ελπίζω να το κάνουν κιόλα. Ε, αν μπορούμε εμεί να διευρύνουμε ή όχι το πεδίο δεν το ξέρω. Πρέπει να το συζητήσω ακόμα με την νομική υπηρεσία, αλλά δεν πρόκανα. Και στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται και από την νομική βάση, ε, καλώς, ε, αν δεν το επιτρέπει η νομική βάση, παρόλα αυτά να βρούμε τρόπο, να δείξουμε και δρόμο ότι για μας είναι σημαντικό να το προχωρήσουμε όσο γίνεται και να το διευρύνουμε, όπως κάναμε και στην τελευταία θητεία. Δυνατότητες πάντα υπάρχουν να το εκφράσεις αυτό, ακόμα και αν δεν υπάρχει νομική βάση και να το συζητήσεις με τα κράτη-μέλη. Και σε ό,τι αφορά την ενισχυμένη συνεργασία, είναι απλή ακρόαση, συναπόφαση εδώ γιοκ. Και γι' αυτό δεν μ' αρέσει Το είπε και η Σόφι Νετβέλτ και στην προηγούμενη θητεία έλεγα και ξανά έλεγα, είχε μαλλιάσει η γλώσσα μου, ότι πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκό δίκαιο. Γιατί είναι το καλύτερο που εξασφαλίζει προστασία για όλα τα κράτη-μέλη. Αλλά δυστυχώς μία χώρα τορπίλησε αυτή την υπόθεση και την οδήγησε σε ένα βάγιο. Υπήρχαν και άλλες χώρες που είχαν πάρα πολύ μεγάλες επιφυλάξεις και ε, άρνηση, πήγα και στις πρωτεύουσε και το συζήτησα, μία χώρα επέμεινε και να βάγισε το εγχείρημα. Τι να κάνουμε, κρίμα. Δεν μπόρεσα εγώ να το αποτρέψω, είπε το κοινοβούλιο στην κυβέρνηση και σε άλλε κυβερνήσει ότι δεν πρόκειται να συμφωνήσει η Βουλή της χώρας, οπότε δεν μπορούμε να πάμε σε ευρωπαϊκό δίκαιο. Ούτε την επόμενη πενταετία σίγουρα. Γι' αυτό ε, είμαστε αναγκασμένοι να ανατρέξουμε σε αυτό το μέσο της ενσημένης συνεργασίας για να περάσει κάτι, εν περιπτώσει. Και οι πολίτες που ενδιαφέρονται στα κράτη που θέλουν να έχουν μια λύση. Οι χώρες που θέλουν να ακολουθήσουν αυτή την ατραπό. Το που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι εξασφαλισμένα τα δικαιώματα των πολιτών μας. Ευχαριστώ. Thank you, Mrs. Ευχαριστούμε. Κυρία Γκέπχαρτ, δεν υπάρχουν ε, άλλα σχόλια. Πάμε στο επόμενο σημείο. Παριθμόν 15. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πακιστάν για την επανεισδοχή. Θα εξετάσουμε το σχέδιο σύστασης. Εισηγητής ο κύριος Όγκορ. Θα σας θυμίσω ότι το Σεπτέμβρη του 2000 ε, έδωσε στην Επιτροπή εντολή το Συμβούλιο για να διαπραγματευτεί συμφωνία με το Πακιστάν για την επανεισδοχή. Έληξαν οι διαπραγματεύσεις το Σεπτέμβριο του 2007 και τέθησε ισχύ το Σεπτέμβριο του 2008 η συμφωνία και το Μάρτιο ε, διαβιβάστηκαν στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο από την Επιτροπή τα σχέδια για την απόφαση που σχετίζεται με αυτή τη συμφωνία. Η κατάσταση έχει αλλάξει πολύ με την ε, συνθήκη της Λισαβόνας. Μετά την ε, Λισαβόνα υπάρχει υποχρεωτική διαβούλευση με το Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του για να υπογραφεί η συμφωνία. Ας ακούσουμε πρώτα τον εισηγητή μας, τον κύριο Σόγκορ, και μετά τους εκπροσώπους της Προεδρίας και της Επιτροπής, αν φυσικά επιθυμούν να παρέμβουν. Και κατόπιν θα ακούσουμε τα μέλη της Επιτροπής. Κύριε Σόγκορ. Ευχαριστώ. Συναντηθήκαμε πριν από ένα μήνα για τελευταία φορά Υπάρχουν δύο βασικά έγγραφα. Το ένα είναι κατά των βασανιστήριων και το άλλο γενικά για θέματα υγείας. Είναι, ε, πρόκειται για μια σύμβαση του ΙΕ το 1994, δεν έχει ολοκληρωθεί η επικύρωση το Πακιστάν δεν είχε αναλάβει ουσιαστικά δέσμευση για την τήρηση αυτών των συμβάσεων. Όταν αρχίσει να ισχύει η συμφωνία περί επανεισδοχής, θα αρχίσουν να ισχύουν και αυτές οι συμβάσεις. Όταν συντάχθηκε αυτό το σχέδιο, δεν είχαμε αυτές τις πληροφορίες στη διάθεσή μας. Άρα θα πρέπει να το αναφέρουμε αυτό στο τέλος του κειμένου. Στην τελευταία παράγραφο έχουμε κάποιες συστάσεις τις οποίες ε, θα σας παρουσιάσω γραπτός. Όταν συζητήσαμε το θέμα αυτό την τελευταία φορά, κάτι το οποίο συζητήσαμε ήταν το γεγονός ότι αν είμαστε βέβαιοι ότι τα άτομα τα οποία θα επανεισαχθούν έχουν παραβιάσει ανθρώπινα δικαιώματα, δεν θα γίνει δεκτή η επανεισδοχή τους. Σε αυτή την περίπτωση βασιζόμαστε στα δικαστήρια των κρατών μελών. Για παράδειγμα, στις 18 Μαΐου είχαμε την εξή είδωση. Αβίτ Νασέρ και Ασμάτ Φαρασκάν, φοιτητές οι οποίοι κατηγορούνται για τρομοκρατία ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, και το δικαστήριο αποφάσισε ότι η επανεισδοχή αυτών των φοιτητών θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο. Γι' αυτό και ακριβώς παρέμειναν στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν ε, ε εστάλησαν στη χώρα τους. Και δεν θα πρέπει φυσικά να λησμονούμε ότι θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και με άλλους τρόπους. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα αυτά θα ε, γίνονται σεβαστά και, στο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις υπόλοιπες χώρες. Ευχαριστούμε. Πριν ακούσουμε τον εκπρόσωπο του, της Προεδρίας και της Επιτροπής, θα ήθελα να δώσω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής, αν τυχόν έχουν να κάνουν ερωτήσεις για αυτό το σχέδιο. Η κυρία Γκυγιώμα. Έχουμε εδώ και καιρό πολλές ερωτη... πολλά ερωτηματικά που έχουν γεννηθεί από προηγούμενες ανταλλαγές απόψεων. Στη συνάντηση δε με την Επιτροπή για τη συμφωνία με το Πακιστάν συζητήθηκαν διάφορα ζητήματα, έγιναν παρατηρήσεις. Ε, δυστυχώς όμως ούτε μέσα στη συμφωνία καλά αυτό αναμενόμενο είναι, αλλά ούτε και στην αιτιολογική έκθεση του εισηγητή δεν υπάρχει ένας απόϊχος, μια καταγραφή όλων αυτών των ερωτημάτων που είχαμε γύρει. Δεν είναι ικανοποιητική η συμφωνία. Αφήστε που σε σχέση με τα ερωτήματα που είχαμε θέσει είναι κάπως ε, γελία η αιτιολογική έκθεση. Θα θέσω πάντως τα ερωτήματα ελπίζοντας ότι θα πάρω κάποιες ε, απαντήσεις. Στην αιτιολογική έκθεση αναφερόμαστε στην αμοιβαιότητα της συμφωνίας. Ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι το θέμα τίθε για την επανεισδοχή προς το Πακιστάν και όχι προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ε, μιλώντας ε, για τους ε, υπηκούς του Πακιστάν και άλλων τρίτων χωρών, κυρίως για τους Αφγανούς ε, κατά ε, πλειοψηφία. Ξέρετε ότι επικρατεί μεγάλη αστάθεια στην περιοχή, οπότε πραγματικά τίθεται ζήτημα ασφάλειας και προστασίας των δικαιωμάτων ε, των ανθρώπων που επιστρέφουν. Τώρα μπορούμε επίσης ε, να αναρωτηθούμε για το εξής. Οι Πακιστανοί οι Αφγανοί που είναι στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μπορεί να ε, θεωρηθεί ότι έχουν μπλοκαριστεί πλέον γιατί έφτασαν πριν τη θέση ισχύ της συμφωνίας και δεύτερον πώς θα καταδειχθεί ότι η ημερομηνία αφήξής τους είναι μεταγενέστερη της υπογραφής της συμφωνίας. μιλάμε επίσης για την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με, από δύο όδους που δεν είναι και συνηθέστερες για να φτάσει κανείς από το Πακιστάν. Ε, και ε, επίσης ε, είπαμε ότι μπορούμε να βασιστούμε στη συμφωνία με την Τουρκία για να σχεδιάσουμε τη συμφωνία με το Πακιστάν, αλλά και εκείνη έχει μπλοκαριστεί. Υπάρχουν και πολλά σαφή σημεία στην ιατολογική έκθεση του εισηγητή η χρήση των ε, σε παραδείγματο χάρη για τι αποχωρήσει, μα δεν συνιστά αυτό λύση σε καμία περίπτωση και σημειώνω επίση ότι ενώ είχαν εκφράσει ανησυχία οι βουλευτές ε, δεν έγινε η αξιολόγηση των συμφωνιών επανεισδοχή ε, που νωρίτερα είχε προσπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με διάφορες άλλε χώρες ή που διαπραγματεύεται ακόμη η Ένωση με άλλες χώρες. Επίσης για τους ανηλίκους δεν αναφέρεται τίποτα για την επανεισδοχή, αλλά δεν αποκλείονται και ρητά από αυτή τη συμφωνία αντίθετα μέσα στο διατακτικό. Το Πακιστάν δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση της Γενέβης, το ξέρουμε, και στην γαλλική εκδοχή είναι προκλητική η διατύπωση, δηλαδή λέμε ότι πρέπει να διαγραφεί αναφορά στη σύμβαση της Γενέβης. Περίεργο μου φαίνεται αυτό. Και επίσης αναφερόμαστε στην απουσία συνοδευτικών μέτρων για τα άτομα που επιστρέφουν. Δεν είναι θαραλέο αυτό το σχέδιο σε σχέση με τις εξουσίες που έχει το Κοινοβούλιο πλέον για την έγκριση διεθνών συμφωνιών, ούτε και απηχεί τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από διάφορα πολιτικά ε, κόμματα για αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε η κυρία Φλότρα. Pour la dynamique du débat, για τη δυναμική της συζήτησης δεν είμαι σίγουρο ότι ήταν καλό που μου δώσατε το λόγο, γιατί η Σιλβί Γκυγιόμ έθεσε εξαιρετικά ερωτήματα. Ε, συμφωνούμε και καλό θα ήταν να απαντήσει η Επιτροπή. Καλό θα ήταν ε, λόγω ε, του ότι υπάρχουν άριθμα ερωτήματα να δώσετε το λόγο στην Επιτροπή για να απαντήσει και να συνεχίσουμε μετά τη συζήτηση. Ας προσθέσω άλλο ένα ερώτημα, αν και δεν πολύ χρειάζεται, γιατί το ανέφερε η Σιλβή. Ε, η προθεσμία, πέρα από τις 30 ημέρες από την υποβολή αιτήματος επανεισδοχής, ε, θεωρούμε ότι γίνεται δεκτή η επανεισδοχή και επικυρώνεται. Ωραία, τι γίνεται με την έκδοση των εγγράφων αν δεν ε, έχουν απαντήσει οι πακιστανικές αρχές. Στις συνεδρίες με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας απάντησαν πως εν τη αυτή περιπτώση μπορούμε να προσφύγουμε στο επωνομαζόμενο Ευρωπαϊκό Λεσέ Πασέ, αλλά είναι μάλλον να ασαφής η νομική βάση του Λεσέ Πασέ. Μπορεί να μας το διευκρινίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάλι. Οι βουλευτές και στα πλαίσια των νέων αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, δεν φαίνεται καλό η Μικτή Επιτροπή Επανεισδοχής να αποκλεί αυτόματα τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίως επειδή υπάρχουν πολλά θέματα παραβία της αρχής της μη επαναπροώθησης, πέρα από τους Αφγανούς που επιτρέπουν στο ε, Πακιστάν ε, και οι Πακιστανοί που στέλνουν τους Αφγανούς στο Αφγανιστάν. στα αρχικά ε, ιστορικά προϊστορικά σχέδια της συμφωνίας, εντάξει καταλαβαίνω ότι δεν το αναφέραμε αυτό, αλλά δεν γίνεται τώρα δεδομένου των νέων αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου να δεχτεί να δεχτούμε την μη συμμετοχή στην Μικτή Επιτροπή και να μην εποπτεύουμε την ε, διαπραγμάτευση της συμφωνίας περί επανεισδοχής. Ο Αντώνιο Γκουτιέρες ε, εδώ στο Κοινοβούλιο δεν ήξερε τι να κάνει, να κλάψει, να γελάσει. Ε, για αυτές τις ε, προσπάθειες, υπέρμετρες προσπάθειες που ισχυρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κάνει συνέχεια για να κλείσει συμφωνία επανεισδοχής, ενώ ε, πολιτικός πως ε, το Πακιστάν είναι η πρώτη χώρα που δεν δέχεται τους πρόσφυγες και άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επανεξετάσει τους όρους επανεισδοχής ε, των Αφγανών προσφύγων που προς το παρόν είναι στο Πακιστάν. Θα πρέπει να είμαστε και λίγο αξιοπρεπείς όταν συζητούμε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ η κυρία Βέμπερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταλαβαίνω και είναι φυσιολογικό να έχουμε ανησυχίες ε, σε σχέση με την ε, Συμφωνία Επανεισδοχής, ε, κυρίως όταν σκεφτόμαστε πώς πόσο δημοκρατική είναι μια χώρα, σε ποιο βαθμό μπορεί να προστατεύσει τα ατομικά δικαιώματα. Ταυτόχρονα όμως πολλά ερωτήματα στα δικά μας τα κράτη-μέλη πρέπει να τα θέσουμε και όχι στο Πακιστάν. Και γιατί αντιτασσόμεθα στη συμφωνία τη αυτή περιπτώσει. Δηλαδή δεν υπάρχει επανεισδοχή εκτό και αν ε, βασιστεί σε μια απόφαση επιστροφή του εν λόγω ατόμου. Οπότε αυτό σημαίνει πω το κράτο μέλο που έχει πάρει την απόφαση πρέπει να ακολουθήσει τις ε, διαδικασίε που σαφώ προσδιορίζονται και περιγράφονται σε διάφορε οδηγίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα όμω ε, πρέπει να συνάδουν και με το διεθνέ δίκαιο που η εφαρμογή του οποίου είναι υποχρεωτική στα κράτη-μέλη μας. Αν διαμένει κάποιος παράνομα, λοιπόν, σε ένα κράτος μέλος, και κατά αυτού έχει ληφθεί απόφαση επιστροφής του, έχει η δικαστική η διοικητική αρχή ε, εξετάσει την υπόθεση αυτή. Μετά ούτε και διεθνή προστασία αυτό το άτομο. Οπότε τι γίνεται ότι μπορεί να δικαστεί σε άλλο επίπεδο η υπόθεση. Αυτό ισχύει όχι μόνο για αυτούς που ενδεχομένως θα επιστρέψουν στο Πακιστάν, αλλά και σε αυτό το, την αρχή του ντόμινο, δηλαδή επιστροφή μέσω μιας χώρας σε άλλη τρίτη χώρα. Οπότε πρέπει να, τα, να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα τα κράτη-μέλη μας. Όταν μας ε, ανησυχεί λέμε ότι μας ανησυχεί η επανεισδοχή στο Πακιστάν, ουσιαστικά μας ανησυχεί το θέμα της επανεισδοχής στα κράτη-μέλη, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Κατά τη γνώμη μου, τι γίνεται τώρα. Όταν έχει ληφθεί απόφαση επιστροφής ε, για κάποιον, διαμένει παράνομα στα κράτη-μέλη της Ένωσης, στα κέντρα κράτησης όσο επιτοπλίστων. Και δεν είναι και το ιδανικό, αυτό που ιδανικά θα θέλαμε να προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε, στη συμφωνία έχουμε την non-affection clause τη ρήτρα που ε, υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να θυγραμμίζονται ε, με την ε, ενωσιακή νομοθεσία και τη διεθνή νομοθεσία περί προστασίας όσων παρανόμως διαμένουν σε κάποια χώρα. Υπάρχει φυσικά η αρχή της μία επαναπρεώθησης. Άρα σε σχέση με τις πακιστανικές αρχές δεν έχουμε και πολλά να πούμε. Στη δική μας επικράτεια πρέπει να βάλουμε τάξη. Ευχαριστώ. Κύριε κυρία Έρνστ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση καταρχήν. Τι κάνουμε εμείς εδώ τώρα. Θέλουμε με μια χώρα ε, να κάνουμε συμφωνία επανειδηστοχής που ξέρουμε ότι δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν τα υπογράφει και ούτε ασχολείται με αυτά που εμείς ε, θέλουμε και κάνουμε. Η βία κατά των γυναικών είναι κάτι τελείως το φυσιολογικό. Είναι καθημερινή δουλειά. Και τα παιδιά από τη ηλικία των 7 ετών μπορούν να διωχθούν και ποινικά. Ε, η ομοφιλοφιλία τιμωρείται έτσι χαλαρά με διετή φυλάκιση. Το λέω κοινικά, αλλά καταλαβαίνετε περί τίνος πρόκειται. Τι συζητάμε, πού είναι η πολιτική και η ηθική μας ευθύνη. Να τα θυμίζουμε και αυτά για να ξέρουμε τι συζητάμε και τι κάνουμε. Αυτό θέλουμε πραγματικά, επανεισδοχή προς τη χώρα αυτή. Και θέλω να ρωτήσω και το Συμβούλιο και την Κομισιόν το εξή. Μια συμφωνία τέτοια επανεισδοχής θα έχει και ε, επιπτώσεις. Θα θεωρηθεί προηγούμενο και θα κάνουμε και άλλες συμφωνίες με άλλες χώρες που περιφρονούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρακαλώ να το σκεφτούμε. Σκεφτείτε τι κάνουμε. Και τώρα έρχομαι σε ερωτήσεις. Το αφγανικό είναι τελείως ανοιχτό. Δεν μου έχει απαντήσει κανένας. Πώς οι Αφγανοί, ας πούμε, που ε, παραδίδονται, ε, που ε, τους επαναδέχονται, πώς θα προστατεύονται και δεν θα τους απελάβουν στο Αφγανιστάν. Τα ξέρουμε αυτά. Τι κάνουμε για όλα αυτά. Γιατί να υποστηρίξουμε μια τέτοια συμφωνία, έστω και κατά διάνοια. Τι γίνεται με τους πολίτες ε, τρίτων κρατών, με τους απάτριδες. λέει ότι θα πρέπει να έχουν φτάσει αεροπορικός. Και ποιες είναι παρακαλώ αυτές οι εθνικότητες, μπορείτε να μου τις πείτε. Με ενδιαφέρει πολύ. Άλλο θέμα. Τα έγγραφα τελείως ασαφής και αόριστη και συγκεχημένη. Ε, τι θα πει ταξιδιωτικά έγγραφα, ποια είναι αυτά. Ε, πολύ απλή ερώτηση. Αυτό το λεγόμενο λεσέ πασέ, το ευρωπαϊκό, η ευρωπαϊκή ταυτότητα, ε, τι είναι αυτό. Η Επιτροπή Επανεισδοχής, τα είπαν οι συνάδελφοι. Μα δεν μπορεί να βγει απ' έξω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να γίνονται αυτά ερήμην του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε τόσο σημαντικά ζητήματα. Ε, τότε τι κάνουμε, γιατί κάνουμε τέτοιες συμφωνίες εμείς. Για την προστασία των δεδομένων, ας μην τα συζητήσουμε καλύτερα. Προστασία των δεδομένων. Εδώ είναι να μην διά τι να σας πω. Σοβαρά τα συζητάμε. Προστασία δεδομένων στο Πακιστάν. Εντάξει, ωραίο. Και μια τελευταία ερώτηση για τη διμερή ε, ε, συμφωνία επανεισδοχής ε, Πακιστάν με άλλες χώρες. Είμαι χωρε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διμερείς ε, συμφωνίες επαναλαμβάνω. Υπάρχουν τέτοιες και αν είναι ποιες. Αυτά. Ευχαριστώ. Η κυρία Νετβέλτ. Στα αγγλικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να ομολογήσω ότι και εγώ δυσκολεύομαι και έχω κάποια ερωτηματικά που πρέπει να μου απαντήσετε πριν με πείσετε. Πρέπει να είμαστε σαφείς εδώ. Δεν συζητάμε την απόφαση που ελήφθη σε κάποια κράτη-μέλη για επανεισδοχή κάποιων Αφγανών στο Αφγανιστάν. Όμως το στοιχείο αυτό έχει σχέση με αυτό που συζητάμε. Διότι την ευθύνη για την απόφαση αυτή και την αξιολόγηση την έχουν τα κράτη-μέλη. Και εμείς υποθέτουμε ότι τα κράτη-μέλη τηρούν την σχετική νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το θέμα είναι, την τηρούν όντω. Εγώ δεν είμαι δικηγόρος, δεν είμαι δικαστής, αλλά αν δω τις αποφάσεις που λαμβάνονται στα κράτη-μέλη για επανειδοχή σε όλες τις χώρες, όχι μόνο στο Αφγανιστάν. Δεν είμαι βέβαιη αν πρέπει να τους επιτευόμαστε στο 100%. Και θα ήθελα λοιπόν κάποιες επιπλέον διασφαλίσεις εδώ. Κάπως να με καθησυχάσετε. Και θα ήθελα να θέσω και μία ερώτηση προς τον εισηγητή, διότι στην τελευταία παράγραφο, στην επεξηγηματική του δήλωση, λέει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν όλες τις ε, σχετικές δράσεις προκειμένου ε, το Αφγανιστάν να κυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση του 1996 για τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα και την Σύμβαση κατά των βασανισμών και άλλων απάνθρωπων ε, συμπεριφορών ή τιμωριών. Εάν είναι σωστή η ανάγνωση που κάνω, οι συζητήσει για τη συμφωνία αυτή γίνονται εδώ και 10 χρόνια, Επομένω, νομίζω ότι το Αφγανιστάν είχε αρκετό χρόνο στη διάθεσή του για να κυρώσει αυτέ τι συμβάσει. Τι μα κάνει λοιπόν να πιστεύουμε ότι αν συμπεριλάβουμε τι συγκεκριμένε ρήτρε τη ε, αποφάση και να του πούμε «Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να τι κυρώσετε αυτέ τι συμβάσει. Ε, Ποιο ο λόγος να το κάνουν τώρα όταν δεν το έχουν κάνει εδώ και 10 χρόνια όταν ε, δεν ενδιαφέρονται από ό,τι φαίνεται να κυρώσουν αυτές τις συμβάσεις. Η επικύρωση των συμβάσεων θα πρέπει να είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ε, ε, συμφωνία αυτή και την υπογραφή της. Ευχαριστώ, κύριε Πουσουτήλ. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ και εγώ με τις ανησυχίες που εξέφρασαν κάποιοι εξημών εδώ και αυτές τις ε, απάνθρωπες εικόνες ε, ανθρώπων που αποστέλλονται στο Αφγανιστάν για να θανατωθούν. Νομίζω ότι το επιχείρημα είναι ε, καθόλου εύλογο και θα ήθελα να με διορθώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν κάνω λάθος, αλλά εγώ το εκλαμβάνω τελείως διαφορετικά το θέμα αυτό. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό. Δεν είναι στόχος αυτής της συμφωνίας αυτό. Η συμφωνία στόχο έχει να αποστείλει στη χώρα τους άτομα τα οποία δεν έχουν καμία... Ε, προστασία, δεν έχουν λάβει καμία δράση προκειμένου να προστατεύονται από τις αρχές μας και από τα δικαστήριά μας. Και μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις, περιπτώσεις στις οποίες δεν δικαιούνται προστασία στην Ευρώπη τα συγκεκριμένα άτομα, θα πρέπει να αποστέλλονται στο Πακιστάν βάσει των όρων αυτής της συμφωνίας. Και νομίζω ότι αυτό είναι το ουσιαστικό σημείο εδώ. Διότι, ιδάλλως, περιπλέκουμε τα πράγματα. Και θα καταψηφίσουμε μια συμφωνία για λανθασμένους λόγους. Και δεν θα πρέπει να καταψηφίσουμε αυτέ τι συμφωνίε ε, για λανθασμένου λόγου. Παρά το γεγονό ότι κατανοώ τα επιχειρήματα τη Σόφη και των άλλων συναδέλφων, θεωρώ ότι εάν δεχτούμε το επιχείρημά σου Σόφη και προχωρήσουμε στο λογικό του συμπέρασμα, τότε σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να κάνουμε καμία συμφωνία επανεισδοχής με καμία χώρα. Διότι πάντα υπάρχουν επιχειρήματα τα οποία λένε ότι τα εθνικά μας δικαστήρια δεν διασφαλίζουν και δεν παρέχουν επαρκή ασφάλεια για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ένα βαθμό τον οποίο εσύ δεν θεωρείς επαρκή. Τα εθνικά δικαστήρια όμως είναι αυτά που λαμβάνουν αποφάσεις και όχι εμείς. Γι' αυτό ακριβώ εξουσιοδοτούμε και τα δικαστήρια να λαμβάνουν αυτέ τι αποφάσει. Θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί εδώ, διότι ουσιαστικά πετάμε και το μωρό μαζί με τα απόνερα και ε, θα καταψηφίσουμε τη συγκεκριμένη συμφωνία για λανθασμένους λόγους. Και η συμφωνία αυτή είναι σημαντική, διότι χωρίς τη συμφωνία το μήνυμα που αποστέλουμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ξέφραγο όλοι. Ε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχει νομοθεσία και οποιοδήποτε δικαιούται προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παραμένει, αλλιώ θα πρέπει να αποστέλλεται στη χώρα του. Πριν ακούσουμε τον εισηγητή, να δώσω δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να μας πει την άποψή του. Κυρίως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνομαι για να μας απαντήσει σε ερωτήσεις που τις ετέθησαν. Ο κύριος Πάλμαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν περάσω σε λεπτομέρειες για τις ερωτήσεις αυτές οι οποίες σας τόθησαν, προς ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο σύστασής του, διότι νομίζω ότι είναι πολύ ισορροπημένη η άποψη που μας παρουσιάζει και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για το έργο του. νομίζω ότι είναι ευπρόσδεκτο από όλη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν γέννη. Ετέθησαν κάποιες ερωτήσεις, κάποιες είναι τεχνικής φύσεως. Θα μπορούσα κάλλιστα να απαντήσω και σε αυτά τα τεχνικά ερωτήματα, αλλά νομίζω ότι ε, θα πρέπει να είναι λίγο πιο διεξοδική η επεξήγηση. Να κάνω όμως κάποιες γενικές παρατηρήσεις καταρχάς. Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις κάποιον από εσά, οι οποίοι λένε ότι θα πρέπει να κάνουμε μια σαφή διάκριση μεταξύ της απόφασης ε, επανεισδοχής και της διαδικασίας επανεισδοχής. Η απόφαση της επιστροφής είναι κάτι το οποίο είναι απόρρια μιας διαδικασίας σε ένα κράτος μέλος για κάποιον ο οποίος δεν διαμένει νομίμως ή ε, δεν ε, εξακολουθεί να διαμένει νομίμως στην χώρα μέλος και στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι δικλείδες ασφαλείας. Και φυσικά, όπως είπε η κυρία Ίνεντβελτ, μπορούμε να αμφισβητήσουμε τις εθνικές αρχές όταν λαμβάνουν τέτοιες αποφάσεις, αλλά δεν νομίζω ότι επαφείται σε εμά εδώ στη συγκεκριμένη αίθουσα και στο συγκεκριμένο κτίριο να αρχίσουμε να αμφισβητούμε τι αποφάσει των κρατών μελών μα. Αυτή είναι μια εντελώ διαφορετική διαδικασία και νομίζω ότι η αρχή την οποία τηρούμε όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι εμπιστευόμαστε τι αρμόδιε αρχέ στο συγκεκριμένο τομέα. Η διαδικασία επανεισδοχή τώρα είναι μια σαφώς διοικητική διαδικασία είναι η φυσική επιστροφή του συγκεκριμένου ατόμου στη χώρα καταγωγής του. Και φυσικά εδώ θα ήθελα να δώσω έμφαση στον όρο καταγωγή, διότι παρά το γεγονός ότι ε, καταρχήν η συμφωνία αυτή προβλέπει και τη δυνατότητα να επιστρέψουν τα άτομα αυτά τα οποία δεν είναι ε, υπήκοοι του Πακιστάν, αν δείτε τις διατάξεις ε, που αφορούν τους ε, υπηκόους τρίτων χωρών, όπως αποκαλούμε, σε καμία περίπτωση μάλλον δεν θα χρησιμοποιηθούν, διότι οι προϋποθέσεις είναι πάρα πολύ αυστηρές. Η διαδικασία λοιπόν επανεισδοχής είναι η διοικητική διαδικασία η οποία επιτρέπει ή διευκολύνει αν θέλετε την επιστροφή κάποιου από μία χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο Πακιστάν σε συγκεκριμένη περίπτωση. Ετέθησαν κάποια ερωτήματα για την αμοιβαιότητα αυτής της συμφωνίας. Στην πράξη φυσικά θα είναι ε, κυρίως υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιβάλλουμε την απόφαση αυτή, τη συμφωνία αυτή στο Πακιστάν. Είναι μια διαδικασία η οποία διήρκησε 5, 6, 7 χρόνια, δεν ξέρω ακριβώς να σας πω, και που επιτρέπει και στο Πακιστάν να απολαμβάνει κάποιον ωφελών. Αν δείτε κάποιες κοινέ δηλώσεις οι οποίες επισυνάπτονται στη συμφωνία θα διαπιστώσετε ότι έχει ε, και κάποιες ε, δυνατότητες νόμιμης μετανάστευσης, πολιτικές για τις θεωρήσεις, ε, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία και επίσης υπήρξαν και πολύ σημαντικές παραχωρήσεις από πλευράς μας στη συμφωνία με το Πακιστάν. Δεν την επιβάλαμε τη συμφωνία αυτή στο Πακιστάν. Το Πακιστάν είναι μια ισχυρή χώρα και σε καμία περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιβάλλει δια της βίας τέτοιες συμφωνίες σε χώρες όπως το Πακιστάν. Κάτι το οποίο αναφέρατε επίση είναι η Κοινή Επιτροπή επανεισδοχή. Η Κοινή Επιτροπή επανεισδοχή δεν προβλέπει τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή αυτή είναι μια τεχνική επιτροπή η οποία παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας. Στην Επιτροπή θα συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη οι επιτροπές αυτές, και εγώ έχω συμμετάσχει σε αρκετές, είναι πολύ τεχνικές και ασχολούνται με τεχνικά θέματα όπως για παράδειγμα την τεκμηρίωση την οποία θα πρέπει να δεχόμαστε επιπλέον των εγγράφων τα οποία συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε με συνεντεύξεις, ε, μιλάμε για πολύ τεχνικές λεπτομέρειες δεν νομίζω ότι το Κοινοβούλιο, το οποίο δεν συμμετέχει στη διαδικασία εφαρμογής αυτής της συμφωνίας, ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε αυτές τις επιτροπές. Με τα χαράς να διαθέσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα ε, συστηματικά τα πρακτικά αυτών των συνεδριάσεων των επιτροπών ε, και με το Πακιστάν αλλά και με άλλες ε, συμφωνίες οι οποίες είναι ήδη ενισχύ. Αλλά το να συμπεριλάβουμε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή την Επιτροπή νομίζω ότι δεν είναι καλή ιδέα. Είχαμε και μια τεχνική ερώτηση για τα ταξιδιωτικά έγγραφα, αν δεν κάνω λάθος. Τι γίνεται με τα ταξιδιωτικά έγγραφα ε, μετά την προθεσμία των 30 ημερών και την εκπνοή τη, Αν δείτε τη συμφωνία, αναφέρομαι στο άρθρο 2, επανεισδοχή υπηκών της χώρας, λέει ότι το ετούν κράτος μέλος θα πρέπει χωρίς καθυστέρηση να δίνει ταξιδιωτικό έγγραφο στον λόγο άτομο, το οποίο έγγραφο θα χρησιμοποιηθεί για την επιστροφή του. Το έγγραφο, από ό,τι λέγεται, θα ισχύει για τουλάχιστον έξι μήνες και αν σε αυτό το διάστημα των 6 μηνών το λόγο άτομο δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει η ε, εγκυρότητα του εγγράφου ε, παρατείνεται για άλλους 4 μήνες. Δεν ξέρω τώρα αν οι ερωτήσεις ε, που κάνατε για το Λεσέ Πασέ ε, ισχύουν εδώ, διότι το Λεσέ Πασέ δεν, προσε... Ε, ε, δεν χρησιμοποιείται σε αυτή τη συμφωνία, δεν προβλέπεται εδώ. Έχουμε ταξιδιωτικά έγγραφα τα οποία θα εκδίδονται και θα έχουν μια ισχύ 6 μηνών και ε, εάν είναι απαραίτητο θα παρατείνεται η εγκυρότητά τους. Να δω λίγο τι άλλο ρωτήσατε. Α, οι Αφγανοί. Η συμφωνία αυτή δεν αφορά την επιστροφή Αφγανών στο Πακιστάν. Μάλιστα, όταν ε, δόθηκε η εντολή αυτή στις αρχές του αιώνα, υπήρχε και ένα πρόγραμμα επανεισδοχής ε, στο Αφγανιστάν, αυτό συμπεριλαμβανόταν και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου να συνεργαστούμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο για ένα πρόγραμμα επιστροφής ε, στο Αφγανιστάν ε, επί βάσεως. Η συμφωνία αυτή κυρίως έχει ως στόχο την επιστροφή των Πακιστανών υπηκόων στη χώρα τους. Βέβαια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμφωνία και για την επιστροφή ενός Αφγανού, εάν ο εν λόγω Αφγανός ε, τηρεί τι προποθέσει που καθορίζονται στο σχετικό άρθρο και φυσικά, επαναλαμβάνω, οι προποθέσει αυτές είναι πάρα πολύ αυστηρέ, διότι ο Αφγανό θα πρέπει στο διαβατήριό του να έχει θεώρηση ή κάποια έγκριση η οποία θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το, ε, εκδοθεί από το Πακιστάν πόσους Αφγανούς έχουμε με έγκυρη θεώρηση ή έγκυρο διαβατήριο ε, με έγκριση η οποία έχει εκδοθεί από τις αρχές του Πακιστάν. Ουσιαστικά λοιπόν αυτή η συμφωνία δεν αφορά Αφγανούς, αλλά αφορά την επιστροφή Πακιστανών υπηκών. Ε, αναφέρθηκε κάπου και η Τουρκία. Ε, έχουμε μεγάλη ροή παράνομων μεταναστών οι οποίοι περνούν από την Τουρκία και φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί εξ αυτών είναι Πακιστανοί. Νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι χρήσιμη αυτή η συμφωνία για να μπορέσουμε να ανακόψουμε αυτέ τι ροέ, διότι αυτό είναι ένα από τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τη σημερινή ημέρα. Τώρα, τι γίνεται με του υπηκόου τρίτων χωρών, ε, ρωτήσατε. Και πάλι αυτό θα μπορούσε να αφορά οποιονδήποτε υπήκο τρίτη χώρας, αρκεί να τηρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στη συμφωνία. Διμερεί συμφωνίε τώρα. Να πω ότι αυτή τη στιγμή όλα τα κράτη-μέλη επιστρέφουν Πακιστανούς υπηκούς στο Πακιστάν. Ακόμα και τούντες άσυλο, τον οποίο η αίτηση έχει απορριφθεί. Τώρα, για διμερεί συμφωνίε επανειδοχή μεταξύ κρατών μελών και του Πακιστάν δεν υπάρχουν τέτοιες συμφωνίε με την εξαίρεση του Ηνωμένου Βασιλείου που έχει ένα μνημόνιο συνενέωση εδώ και ένα-δυο χρόνια αλλά οι υπόλοιπε χώρε δεν έχουν διμερείς διευθετήσει ή συμφωνίε με ε, το Πακιστάν. Νομίζω ότι απάντησα τις περισσότερες από τις ερωτήσεις σας, αν έχει όλες. Ε, μπορώ κάλλιστα να απαντήσω και σε άλλες ερωτήσεις, αν υπάρχει χρόνος ή ανάγκη για να απαντήσω. Προς τα παρόν θα σιωπήσω. Ευχαριστώ. Mr. Now for the presidency, Senor Burgos. Ο κύριος Μπούργος, από την Προεδρία. Ε, buenos días. Καλημέρα σας. Δεν είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε εδώ να συζητήσουμε για τη συμφωνία επανεισδοχής με το Πακιστάν. Ακούσαμε προσεκτικά και τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας και ήθελα να σας πω ότι για το Συμβούλιο η συμφωνία αυτή έχει τεράστια σημασία. Οι συμφωνίες επανεισδοχής είναι βασικό συστατικό της πολιτικής μετανάστευσης των κρατών μελών και τώρα λογικά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν δεν υπογραφεί η κοινοτική συμφωνία, μπορούν τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε διμερείς συμφωνίες. Αλλά βεβαίως και λογικά με πολύ περισσότερες δυσκολίες από εκείνες που αντιμετωπίζουμε όταν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέχεται και αναλαμβάνει τις ευθύνες της στην ε, πολιτική μετανάστευση. Συγκεκριμένα τώρα, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία με το Πακιστάν, δώσαμε εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματευτεί και με μεγάλη ικανοποίηση δεχτήκαμε το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, το γνωρίζουμε αυτό, αλλά το τελικό αποτέλεσμα πιστεύουμε ότι είναι πολύ ε, λογικό και το υποστηρίζουμε. Επίσης, για τον ίδιο λόγο, συμφωνώ με την απάντηση που μόλις έδωσε ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις οποίες απαντήσεις σε όλα τα θέματα προσυπογράφουμε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικά θέματα, γιατί βλέπω ότι σας ανησυχούν. Ε, τους βολευτές εδώ. Πρώτον, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι προφανές ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουμε δεσμευθεί και είμαστε προσιλωμένοι στην υποχρέωση που έχουμε να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα όμως να τονίσω ότι στη Συμφωνία Επανεισδοχής περί τίνος πρόκειται. Είναι μια συμφωνία που έρχεται όταν έχουν γίνει όλες οι εξακριβώσεις. Δηλαδή, αν έχει δικαίωμα σε διεθνή προστασία, ε, ότι δεν διώκεται, ότι δεν υπάρχει αρχή της μη επαναπροώθησης. ρεφουλμό. Και από εκεί και πέρα ε, εκδίδεται το ένταλμα απέλασης και επανεισδοχής και είναι η τελευταία φάση δηλαδή, εφόσον έχουν εξαντληθεί όλα τα στάδια και έχει επαληθευθεί και έχει ξεκριβωθεί ότι το πρόσωπο αυτό δεν κινδυνεύει να παραβιαστούν τα ανθρώπινα του δικαιώματα επαναπροωθούμενο. Ένα άλλο θέμα που σας ανησυχεί πολύ από ό,τι είδα είναι οι, πίκο, οι πολίτες τρίτων χωρών. βασικός στόχος, ξέρετε, είναι η επαναπροώθηση Πακιστανών πολιτών, έτσι ε, όχι τρίτων χωρών. Και αυτό θεωρούμε ότι θα συμβεί ε, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων. Σε ό,τι αφορά τώρα πολίτες τρίτων χωρών συμπεριλαμβανομένων και των Αφγανών, θα είναι έκτακτες ε, περιπτώσεις αυτές και εξαιρετικές και το ορίζει και η συμφωνία πότε μπορούν να επαναπροωθούνται σε περίπτωση που θα έχουν ένα ταξιδιωτικό έγγραφο που θα έχει εκδώσει το Πακιστάν, είτε βίζα, θεώρηση διαβατηρίου, είτε άδεια ε, διαμονής ή έρχονται από το Πακιστάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τρόπο λαθρέο και παράνομο. Βέβαια αυτό είναι η απόλυτη εξαίρεση αν σκεφτεί κανείς πόσο μακριά είναι η χώρα αυτή. Δηλαδή κάποια σχέση θα έχουν με το Πακιστάν για να επαναπροωθηθούν στο Πακιστάν οι άνθρωποι αυτοί. Και βεβαίως ισχύουν πάντα οι ίδιες προφυλάξεις και τα μέτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν πρόκειται να επαναπροωθηθεί κανείς στο Πακιστάν αν δεν είναι βέβαια το κράτος μέλος ότι θα γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματά του. Και αρχή της μη επαναπροώθησης ισχύει, το non που λέμε. Αυτά. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ε, παρακαλέσω να καταλάβετε πόσο σημαντική είναι η υπογραφή αυτής της συμφωνίας και να εκφράσω ότι συμφωνούμε με την έκθεση του εισηγητού. Ευχαριστώ πολύ. Now back to you, Mr. Sogor, if you want to react. Κύριε Σόγκορ, τώρα θα σας ξαναδώσουμε το λόγο μήπως θέλετε να απαντήσετε σε όλα αυτά τα σχολεία και να σχολιάσετε και τις απαντήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τις ερωτήσεις που υπευλήθησαν από τα μέλη της Επιτροπής για το νομικό καθεστώς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω συναδελφούς Βέμπερ και Μπουσουτήλ για τα σχόλιά σας, καθώς επίσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Δεν θα απαντήσω σε όλα. Επιτρέψτε μου όμως να απαντήσω στην κυρία Ινετβέλτ πρώτα απ' όλα. Μάλλον δεν έχουμε καταλάβει κάτι. Οι συμβάσει αυτές έχουν κυρωθεί από τη Βουλή του Πακιστάν. Και προηγουμένως μιλήσαμε και για την εμπιστοσύνη απέναντι στις δικαστικές αποφάσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν επαναπροώθησε τους πολίτες για, αυτούς γιατί ήξερε ε, ότι δεν μπορεί να είναι σίγουρο ότι θα εφαρμοστούν ε, από το κράτος αυτά που πρέπει ως εγγύησης. Εγώ προέρχομαι από την Ανατολική Ευρώπη που δεν είχαμε μεγάλη εμπιστοσύνη στο κράτος, ε, αλλά νομίζω ότι ε, η δικαιοσύνη είναι αξιόπιστη, μη τι άλλο στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιο σκιώδη ηγητή μίλησε για αναδρομική ισχύ. Δεν πρόκειται για αναδρομική ισχύ. Ε, για αμοιβαιότητα πρόκειται για αμοιβαία ε, αναγνώριση και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τέτοιων ε, ζητημάτων. Δηλαδή, μπορεί σε κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, να έχουμε παραβιάσεις και καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην Ένωση. Ακόμα χειρότερες από αυτές που ενδεχομένως να συμβαίνουν στο Πακιστάν. Παρένθεση αυτή. Προσωπική μου άποψη είναι. Όχι η άποψη ε, του κόμματος το οποίο εκπροσωπώ και της πολιτικής μου ομάδας. Εν περιπτώσει, για το μέλλον, πρέπει να σας πω ότι ορισμένα κείμενα έχουν ήδη λήξει, έχουν τελειώσει, έχουν υπογραφεί, δεν μπορούμε να τα τροποποιήσουμε, αλλιώς θα χρειαστεί τροποποίηση της συνθήκης ποια είναι λοιπόν η σύσταση δική μου ως εισηγητού και θέλω να το πω και σε όλες τις πολιτικές ομάδες και σε όλους τους ε, σκιώδεις εισηγητές γιατί θα συνεδριάσουμε τον Ιούνιο ε, να τα ξαναπούμε τότε στην Ολομέλεια του Ιουνίου που έχουμε τη νέα συνεδρίαση για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Άρα λοιπόν θα δοθεί συνέχεια και θα έρθετε σε επαφή, όπως λέτε, με τους σκιώτης ηγητές για να συζητήσετε μαζί τους τα επόμενα βήματα. Ισχύει αυτό? Ωραία. Έστω λοιπόν, ε, ολοκληρώνεται και αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης και πάμε στο επόμενο, που είναι το 16. Πολύ σημαντικό επίσης. Ακρόαση θα τη χαρακτηρίζα παρουσίαση ε, της ετήσιας έκθεσης της Eurojust έχουμε ε, τον πρόεδρο της Eurojust ενώπιόν μας. Τον καλωσορίζουμε θερμότατα. Καλώς ορίστε κύριε Williams. Καθίστε παρακαλώ. Good to see you. We welcome Mr. Alec Καλωσορίζουμε τον κύριο Άλετ Βίλιαμς, πρόεδρο της Eurojust. Για τα τελευταία 35 λεπτά τη σημερινή συνεδρίασης της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ τον ακούσαμε το Μάρτιο πρώτη φορά. Τιμήσε με την παρουσία του την ε, Επιτροπή μας. Ε, μας έκανε μια πρώτη παρουσίαση. Όργανα όπως η Eurojust είναι το κομμάτι των μελλοντικών εξελίξεων στο χώρο ε, ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Συστάθηκε το 2002 η Eurojust. Έκτοτε έχουν ε, σημειωθεί πολλές εξελίξεις. επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα του οργανισμού αυτού από αυτές τις εξελίξεις. Η ετήσια έκθεση του 2009 της Eurojust έχει σημαντικά στοιχεία. Θα ακούσουμε την παρουσίαση του Προέδρου. Κατόπιν θα γίνει η συζήτηση. Μετά τις παρουσιάσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε για τα καλά σας λόγια και για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω την ετήσια έκθεση για το 2009 της Eurojust στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. 10-15 λεπτά έχω στη διάθεσή μου, έτσι. 10, ε. 10. Ευχαριστώ. Έχω επίγνωση του ότι εφόσον ε, είχα την ευκαιρία να σας μιλήσω το Μάρτιο μπορεί να έχετε μια αίσθηση ντεζαβή, να τα έχετε ξανακούσει, να έχετε μια αίσθηση ότι έχετε ξανακούσει αυτά που σας λέω, αλλά... Μην ξεχνάμε ότι το 2009 υπήρξαν δύο σημαντικές εξελίξεις ε, στη Eurojust, ε, δηλαδή η μονάδα της δικαστικής συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρώτη εξέλιξη προφανής και βαρύνουσα είναι το, τοπικό, το νομικό τοπίο συγγνώμη, της Eurojust μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, ε, τη δημοσίευση του προγράμματος της Στοκχόλμης. Και για μας ε, κάτι άλλο πολύ σημαντικό, η έκδοση της ε, απόφασης της Eurojust. Δεύτερον, σε αυτή τη σύντομη παρουσίαση θα σας μιλήσω για τις ε, αλλαγές ε, της ίδιας ε, της ετήσιας έκθεσης μετά από συστάσεις που λάβαμε αντιλαμβάνουμε ότι έχετε λάβει τουλάχιστον στα αγγλικά την ετήσια έκθεση τη Eurojust. Εν πάση περιπτώσει, ταχύτατα θα υπάρχει σε όλες τι επίσημε γλώσσες αυτή η ετήσια έκθεση. Πρέπει να εστιαστούμε λοιπόν στι τρέχουσε εργασίε και στα εμπόδια ε, τη δικαστική συνεργασία σε ποινικέ υποθέσει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αρχίσω με κάποιε σύντομε παρατηρήσει ε, για τις ε, σχέσει ανάμεσα στη Eurojust και την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Είναι η πρώτη έκθεση που παρουσιάζεται μετά τη θέση ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα, όπω σα έλεγα. Πρώτη παρατήρηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αρμοδιότητες για την αξιολόγηση της Eurojust, άρθρο 85 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί σαφώς προβλέπεται ότι όταν ε, προκύψει ο κανονισμός της Eurojust και εκτιμάται ότι γύρω στο 2012 θα ε, θεσπιστεί ο κανονισμός, τότε το Κοινοβούλιο θα εμπλακεί στην αξιολόγηση της Eurojust. Δεύτερη παρατήρηση για αυτό το θέμα. Έχουν γίνει ήδη βήματα, ούτω ώστε η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών να εμπλακεί ήδη στην αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της Eurojust. Αναμένεται σύντομα επίσκεψη από μέλη της Επιτροπής σας ε, στη Eurojust στις 29 Ιουνίου μάλιστα. Εκπρόσωποι της Επιτροπής σας ε, θα μεταβούν ε, στη Eurojust για να συμμετάσχουν σε μια ε, συνεδρία που ονομάζεται Άτυπη Ομάδα Εργασίας και ασχολείται με την υλοποίηση και εφαρμογή των διατάξεων της νέας απόφασης Eurojust από πλευράς των κρατών μελών. Ελπίζουμε ότι τα θέματα που θα συζητηθούν σε αυτή τη συνεδρίαση θα παρουσιάσουν ενδιαφέρον για τα μέλη της Επιτροπής σας. Ε, τρίτη ε, προκατακτική ε, παρατήρηση, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών δεδομένων των αρμοδιοτήτων που έχει για την απαλλαγή του προϋπολογισμού της Eurojust έχει ήδη δηλώσει ότι αυτή η απαλλαγή ενέχει και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της Eurojust. Οπότε γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι δουλειά του Κοινοβουλίου για όλα αυτά τα ζητήματα. Πολύ σύντομα τώρα θα ήθελα να σας μιλήσω για τους φακέλους που χειρίζεται η Eurojust, δηλαδή το μεγαλύτερο όγκο της αιτήσιας έκθεσης και τις ανησυχίες που υπάρχουν και προκύπτουν μέσα στην έκθεση. Το πρώτο θέμα είναι ότι τα κράτη-μέλη συνεχίσουν να κάνουν καταγγελίες για διάφορες, ε, να παραπέμπουν συγγνώμη, διάφορες υποθέσεις στη Eurojust ε, τα τελευταία 8-9 χρόνια από την ε, σύσταση της Eurojust και μετά από το 2002. Ε, πλασιάστηκαν οι υποθέσεις που παραπέμπονται στην Eurojust και η αύξηση κλιμακώνεται κάθε χρόνο. Δείτε για το 2009 τα αριθμητικά στοιχεία. Αν ε, τα συγκρίνετε με το 2008 θα δείτε ότι σημειώθηκε αύξηση 15% στον αριθμό των περιπτώσεων που ε, παραπέμπονται στην Eurojust και καταγράφονται στο δικό μας σύστημα. Τώρα χειριζόμαστε 14.000 περίπου υποθέσεις το χρόνο ε, συγγνώμη, 1.400 υποθέσει το χρόνο. Και οι χώρες ε, όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Πολωνία ε, είναι οι χώρες που μας προτιμούν, που μας χρησιμοποιούν περισσότερο. Τα στοιχεία προέκυψαν χτες ε, και δείχνουν ότι τους πρώτους πέντε μήνες του 2010 Ε, καταγράψαμε 600 περίπου υποθέσεις στο σύστημά μας. Άλλα βασικά ζητήματα ε, του, του έργου της Eurojust είναι ε, πρώτον οι, συνε, οι συντονιστικές συνεδριάσεις. Πέρσι έγιναν 131 τέτοιες συντονιστικές συνεδριάσεις στη Eurojust ε, και αυτό δείχνει την προστιθέμενη αξία μας στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας. Τι γίνεται σε αυτές τις συντονιστικές συνεδριάσεις. Έχουμε έναν εισαγγελέα και έναν ανακριτή, ένα δικαστή του κράτους μέλους που εμπλέκεται στην υπόθεση που έρχεται στη Eurojust Κάθεται λοιπόν σε ένα τραπέζι και συζητάει την υπόθεση, την τακτική που ακολουθείται στην ε, συγκεκριμένη υπόθεση, ρυθμίζει ε, ιδιαίτερες δυσκολίες όταν υπάρχει σύγκρουση αρμοδιοτήτων, ε, το θέμα του χρονισμού των εκτελεστικών πράξεων σε κάθε κράτος μέλος. Έτσι καταλαβαίνετε, Βερτίνος πρόκειται. Σας είπα ότι έχουν γίνει 131 τέτοιε συντονιστικέ συνεδριάσεις πέρσι και τα δύο τρίτα αυτών των συνεδριάσεων αφορούσαν σε περισσότερα από τρία κράτη-μέλη. Κάτι άλλο ενθαρρυντικό κατ' εμέ είναι ότι από αυτές τις 131 συνεδριάσεις είχαμε σημαντική συμμετοχή της Europol, ε, τους ε, ε, γείτονές μας δηλαδή στη Χάγη. Στις 47 υποθέσεις συμμετείχε και η Europol, στο 1 τρίτο περίπου δηλαδή. Και πάλι υπάρχει παρεμφερή στάση για το 2010. Στους 5 μήνες που έλεξαν χτες είχαμε 61 συντονιστικές συνεδριάσεις στη Χάγη. Ένα τελευταίο σημείο για αυτές τις γιατί γενικότερα για τις δραστηριότητές μας είναι το εξής. Η Eurojust έχει ρόλο στις κοινέ ερευνητικέ ομάδες. Υπάρχουν δύο πτυχές σε αυτό το ζήτημα. Πρώτον, η Eurojust θα είναι το κέντρο για το δίκτυο των κοινών ερευνητικών ομάδων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεύτερον ε, έχει ενεργό ρόλο η Eurojust ε, στη διοικητική χρηματοδότηση που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτές τις κοινέ ερευνητικέ ομάδες. Πέρσι ε, πήραμε κονδύλια πρώτη φορά, δηλαδή για να τα διαχειριστούμε εμείς έτσι, για τις κοινέ ερευνητικέ ομάδες. Με επιτυχία το διαταχειριστήκαμε. Ε, στα τέλη του 2009 έφτασαν τα κονδύλια και πέντε ερευνητικές ομάδες πήραν τέτοια χρηματοδότηση υπό την αιγίδα της Eurojust. Και επειδή με επιτυχία διαχειριστήκαμε αυτή την χρηματοδότηση και την επιχειρησιακή λειτουργία των κοινών ερευνητικών ομάδων, δέχτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρουμε περίπου 2,1 εκατομμύρια ευρώ για περαιτέρω διαχείριση των κονδυλίων για αυτές τις ε, κοινέ ερευνητικέ ομάδες. Επίσης, συνεργαστήκαμε με την Europol για την εκπόνηση εγχειριδίου για τις κοινέ ερευνητικέ ομάδε ε, με στόχο κυρίω ε, για του ερευνητέ ανακριτέ εισαγγελεί, τέλο πάντων για του επαγγελματίε ε, του τομέα αυτού ή στα κράτη-μέλη και υπάρχει αυτό το εγχειρίδιο σε όλε τι επίσημε γλώσσε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, υπερεύει ήδη το χρόνο μου, Πρόεδρε, δεν είμαι σίγουρο. Όχι, ωραία. υπάρχει ένα άλλο θέμα που καλό είναι να το συζητήσουμε εν συντομία γιατί μετά την περσινή ετήσια έκθεση μας το ζήτησαν να εντοπίσουμε τις ε, δυσκολίες που αντιμετωπίζει η δικαστική συνεργασία. Όταν ε, δείτε την έκθεση θα συνειδητοποιήσετε ότι υπάρχουν δύο βασικές ομάδες δυσκολιών έτσι, που εντοπίζονται. Πρώτη ομάδα, οι πρακτικές δυσκολίες, έτσι τις ονομάζουμε εξυπακούεται ότι πάντοτε θα υπάρχει θέμα, ε, πρόβλημα πόρων έτσι, για την καταπολέμηση του εγκλήματος και κυρίως της διασυνοριακής εγκληματικότητας. Πέραν αυτού όμως ε, υπάρχει θέμα ε, του, της διασυνοριακής εγκληματικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι το ονομάσαμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει μια συμμορία οργανωμένου εγκλήματος σε ένα κράτος μέλος και ε, στοχεύει θύματα σε άλλο κράτος μέλος ή εν λόγω συμμορία. Προφανώς θα προκύψουν δυσκολίες για να ερευνήσουμε και να διώξουμε αποτελεσματικά τα εγκλήματα. Και οι δυσκολίες αυτές μπορεί να είναι τεχνικού χαρακτήρα. Δηλαδή υπάρχουν, ε, υπάρχει θέμα δικαιοδοσίας. Ε, η ομάδα οργανωμένου εγκλήματος στο κράτος μέλος Α έχει μια δραστηριότητα που ε, δεν χαρακτηρίζεται ως εγκληματική βάσει της νομοθεσίας του κράτους μέλους Α. Οπότε, στην πράξη είναι πάρα πολύ δύσκολο να χαρακτηρίσουμε αυτή την αξιόπινη πράξη. Ε, αν οι δραστηριότητες ε, του κράτους μέλους Α όμως, που ξεκινούν από το κράτος μέλους Α, διεξάγονται στο κράτος μέλος Β, τότε δημιουργούνται δυσκολίες αν προκύψει απόφαση από το κράτος μέλους Β. Και η απόφαση του κράτους μέλους Β θα επηρεαστεί από αυτή την κατάσταση. Ξαναλέω, αν οι εγκληματίε του, του κράτου Α στοχεύουν θύματα στο κράτο Β, έχουμε πρόβλημα με τον χαρακτηρισμό τη αξιόπινη πράξη. Και βλέπετε στι δραστηριότητε μα ε, από την τήσια έκθεση ε, ότι ε, δυσκολευόμαστε με, σε θέματα συνοριακής απάτης, όπως το, τα αποκαλούμε, border front. Επίσης υπάρχουν νομικά, πολιτιστικά ζητήματα που μας δυσκολεύουν και ε, είναι ε, ε, πολυσχηδές το πρόβλημα. Αυτό τι σημαίνει, έχουμε διαφορετικά ένομα συστήματα, διαφορετικούς ρόλους για ένα δικαστή, για έναν εισαγγελέα, για έναν ανακριτή. Ένα παράδειγμα, η έγκριση για μια ελεγχόμενη παράδοση. Σε ένα κράτος μέλος μπορεί να είναι θέμα δικαστή, έτσι, ή ένα, ανακριτή. Σε άλλο κράτος μέλος μπορεί να είναι καθαρά αστυνομική δραστηριότητα να εγκριθεί μια ελεγχόμενη παραλαβή. Άμα όμως μία ελεγχομένη παραλαβή ε, καλύπτει ή περισσότερα κράτη-μέλη, διασχίζει τα σύνορα, υπάρχει πρόβλημα για την ε, χορήγηση της έγκρισης. Ε, δηλαδή, ποιο είδους μέσα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε δύναμη της νομοθεσίας της Ένωσης. Προφανώς προκύπτουν και δυσκολίες για το παραδεκτό των τεκμηρίων, των αποδεικτικών στοιχείων. Πρόεδρε, ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο. Καλό θα ήταν να το αφήσω αυτό το θέμα. Ε, τώρα, ένα συμπέρασμα. Υπάρχουν κομμάτια μέσα στην έκθεση που αναφέρονται στους εταίρους μας, σε επίπεδο ένωσης δηλαδή. Θα ήθελα να αναφερθώ πρώτον το, στο Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο, είναι βασικός εταίρος της Eurojust και ελπίζουμε ότι μετά τη συνεδρία 29 Ιουνίου όπου φυσικά προσκαλούμε την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, θα προκύψουν και άλλες πρωτοβουλίες ε, για να αναπτυχθεί η σχέση και το μοίρασμα των εργασιών ανάμεσα στη Eurojust και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και θα αναβαθμιστεί η συνεργασία μας. Άλλος βασικός εταίρος είναι η Europol και πέρσι ε, σημειώθηκε σημαντικότατη πρόοδος ε, γιατί υπογράψαμε νέα συμφωνία συνεργασίας με τη Europol χάρη στην οποία θα υπάρξει καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στους δύο οργανισμούς νωρίτερα η ανταλλαγή αλλαγή είχε περιγραφεί ως ότι γίνεται μόνο όταν είναι απαραίτητη. Τώρα όλα έχουν γίνει πολύ πιο συγκεκριμένα και ελπίζουν να ενεργοποιηθεί η ανταλλαγή ε, πληροφοριών με αυτή τη νέα συμφωνία συνεργασίας. Όπως σας είπα, η Europol ε, παρευρίσκεται στις συντονιστικές συνεδριάσεις μας και έχουν αρχίσει να μας ε, μιμούνται, να το πω έτσι κολακεύοντας τη Eurojust, μιμούμε, Εκτιμούνται λοιπόν τον τρόπο εργασίας μας ε, και 12 από τις 19 ε, υποθέσεις ε, ανάλυσης ακολούθησαν αυτή τη διαδικασία. Ένα τελευταίο παράδειγμα. Κάτι στις δραστηριότητες της Eurojust που δεν προκύπτει μέσα στην ετήσια έκθεση, αλλά προκύπτει από μία υπόθεση που ανέλαβε από κοινού η Eurojust και η Europol πριν από λίγες εβδομάδες είναι η υπόθεση χρηματοδότησης μιας Ισλαμικής τρομοκρατικής ομάδας, ενδιαφέρουσα υπόθεση κατά με, άρχισε στην Ιταλία ε, και είναι ξεκάθαρο ότι η χρηματοδότηση των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων έγινε ε, μέσω δραστηριο... εμπορίας ε, ανθρώπων, κυρίως ε, στην Ινδική Χερσόνησο και με... από εμπόριο ναρκωτικών επίσης. Η Eurojust πλάκη σε μεγάλο βαθμό σε αυτή την υπόθεση. Έγιναν συντονιστικές συνεδριάσεις στην έδρα μας και τελικά ξεδόθηκαν ε, εκδώσαμε εντάλματα συλληψή ε, και πέντε συνελήφθησαν που είχαν συμμετάσχει στη χρηματοδότηση αυτών των ε, δραστηριοτήτων. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση, σας ευχαριστούμε που μας βοηθήσετε να συζητήσουμε το θέμα αυτό και να έχουμε λίγο χρόνο να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη της Επιτροπής μας. Βλέπετε εδώ πέρα και την έντυπη έκδοση της ετήσιας έκθεσης της Eurojust. Είναι στη διάθεση των μελών για να έχουν μια πλήρη ανάλυση του έργου της Eurojust ε, στη διάρκεια του 2009. Να ακούσουμε τώρα τους ε, συναδέλφους. Ο κύριος Λαμπρινίδης καταρχάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίσατε κύριε Williams. Η ερώτησή μου σχετίζεται με το παράδειγμα που παρουσιάσατε στο τέλος, το SWIFT και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Όπως θα γνωρίζετε, το βασικό θέμα κατά τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας ε, SWIFT λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να εξετάσει αιτήματα των Ηνωμένων Πολιτειών για την αποδέσμευση πληροφοριών SWIFT και την ε, δυνατότητα να τις δουν επί τη βάση στοιχείων που παρουσιάζονται για γνωστούς σε αυτούς υπόπτους τρομοκρατίας. Η ερώτησή μου προς εσάς είναι η εξής. Πώς μπορεί η Eurojust και τι εξουσιοδότηση πέραν αυτής που ήδη διαθέτει θα χρειάζεται προκειμένου να μπορέσει, εάν προκύψει και τέτοια ανάγκη, να διαδραματίσει αυτό το ρόλο ε, στα πλαίσια και της ε, ένταξης της στη συνθήκη της Λισαβόνας. Ευχαριστώ, κυρία Βέμπερ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τον κύριο Βίλιαμς για την παρουσίασή του και καλή τύχη στο έργο σας. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο περισσότερα πράγματα για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει Eurojust. Ε, ε, με ικανοποιούν τα θετικά στοιχεία και ξέρω ότι δεν ήταν εύκολο ακόμα και το να πιέσετε για κάποιες από τις αλλαγές που τελικά έγιναν αποδεκτές. Αλλά επειδή θα θέλαμε να σας δώσουμε και περισσότερες εξουσίες στο μέλλον, θα ήθελα να ακούσω κάποια περισσότερα πράγματα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, ώστε να μπορέσουμε να τα επιλύσουμε. Και όταν ε, λέω προβλήματα, αναφέρομαι για παράδειγμα και ε, στις κοινέ ομάδες έρευνας, ε, την, το δισταγμό που υπάρχει από πλευράς κρατών μελών σε κάποιες περιπτώσεις. Αναφερθήκατε και σε κάποιες δυσκολίες και είπατε ότι υπάρχουν και διαφορετικά νομικά συστήματα και διαφορετικές συνήθειες από νομικής πλευράς. Ε, θα ήθελα να ακούσω περισσότερα για παραδείγματα που όπως ε, μας είπατε στο τέλος της παρουσίασης και πώς ασχολείστε κατά βάση με τα θέματα αυτά όταν ε, πρέπει να τα αντιμετωπίσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ιακολίνο. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βίλιαμς, άκουσα πολύ προσεκτικά όλα όσα μας αναπτύξατε και όλα όσα είπατε για τις δραστηριότητες στις οποίες αναφερθήκατε. Στο 4 βγαίνουν τα αγγλικά, λέει ο κύριος Ιακολίνο. Το 2 είναι για τα αγγλικά. Το βρήκαμε. <laughs> Ακούσαμε λοιπόν πολύ προσεκτικά τα στοιχεία τα οποία μας δώσετε, 700 υποθέσεις ε, τους τελευταίους πέντε μήνες, μεγαλύτερο συντονισμό, 131 συνεδριάσεις, ε, ε, μια συμφωνία συνεργασίας με τη Europol, κοινέ ομάδες έρευνας, οικονομική πόροι που διατίθενται προς αυτό το σκοπό. Μεγάλη κινητικότητα λοιπόν από πλευράς Eurojust. Η ερώτησή μου είναι πάρα πολύ απλή. Σήμερα ασχοληθήκαμε πιο επισταμένα με το θέμα της Ευρωπαϊκής Εντολής Προστασίας. Ε, μία εντολή η οποία απαιτεί προστασία και συνεργασία μεταξύ ε, κρατών μελών. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Η συμμετέχει σε προληπτική εντό εισαγωγών συνεργασία, ώστε τα θέματα τα οποία συζητούνται και καθορίζονται πρώτα στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και στη συνέχεια στην Ολομέλεια συνάδουν με την αποστολή της Eurojust. Διότι αυτό που έχει σημασία είναι το νομοθετικό πλαίσιο να είναι συνεκτικό με τους στόχους που θέτει αυτή η δομή και οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να υλοποιούνται και μέσω της συνδρομής σας, ε, από τεχνικής πλευράς φυσικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άλλες ερωτήσεις. Ναι, ο κύριος Μπρόνς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης θα χρησιμοποιηθεί για να εκδίδεται κάποιος από μια χώρα που αυτό που έχει κάνει δεν είναι αδίκημα σε άλλη χώρα που είναι αδίκημα. Αυτό αφορά ε, ε ας πούμε μια ερετική άποψη ε, ακαδημαϊκή ή πολιτική. Γιατί υπάρχουν κάποιες χώρες που το θεωρούν αυτό έγκλημα πολέμου, ενώ κάποιες άλλες επιτρέπουν να τα λες αυτά τα πράγματα. Κύριε Δίας μέρα θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλές ερωτήσεις έχω εγώ, αλλά για λόγους χρονικούς θα κάνω μία μόνο. Ευχαριστώ, ε, κύριε Williams. Σε ό,τι αφορά τις συντονιστικές αυτές συνεδριάσεις, συγκεκριμένα ε, όταν υπάρχει διένεξη ε, δικαιοδοσίας, θα ήθελα να μου πείτε ποιοι συμμετέχουν εκεί, ποιοι ενέχονται είναι το κράτος μέλος, είναι ο αρμόδιος δικαστής. Στην περίπτωση της Ισπανίας είναι το ανώτατο δικαστήριο, είναι η Audiência Nacional, το δικαστήριο για ε, ε, την τρομοκρατία. Ε, είναι ένας πρωτοδίκης. Ποιος συμμετέχει εκεί στις συντονιστικές αυτές προσπάθειες όταν έχουμε πρόβλημα δικαιοδοσίας. Μάλιστα. Πριν επανέλθει ο κύριος Williams αν θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Προεδρία να μιλήσει, το Συμβούλιο, αν παρευρίσκονται. Όχι, όχι. Δεν βλέπω τέτοιου εκπροσώπου εδώ, ούτε Συμβούλιο. Εσεί έχετε το λόγο τώρα, κύριε Βίλιαμ, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα στι απαντήσει μου να επανέλθω στα ερωτήματα. Ε, πρώτα του κυρίου Λαμπρινίδη για το SWIFT Η ε, Eurojust παίρνει ε, πληροφορίες ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό, ενημερώνεται από τα κρατη δηλαδή. Ο ρόλος μας είναι να ενισχύουμε και να υποστηρίζουμε τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών διοκτικών αρχών και της εισαγγελία. Αυτό το λέει και η συνθήκη δηλαδή, έτσι ορίζει το ρόλο μας. Μπορεί λοιπόν να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες η Eurojust ε, αλλά μπορούν να προσφεύγουν σε μας και άλλοι εκτός από τις διοκτικές αρχές και την εισαγγελία. Ακριβώς επειδή έχουμε σχέση και με την ε, Europol το λέω αυτό. Ε, δηλαδή μπορεί και εκείνοι να προσφεύγουν. Αυτό το λέω εισαγωγικά και θα έρθω και στην ερώτησή σας ε, για ε, τις πληροφορίες λοιπόν που λαμβάνουμε. Ποιες είναι. Είναι και προς όφελος των διοκτικών αρχών και βεβαίως παραμένουν και ε, κύριοι της πληροφορίας ε, και αν ε, χρειαστεί και περαιτέρω διαβίβαση της πληροφορίας αυτής, η Eurojust είναι υποχρεωμένη να ρωτάει τις αρχές αν μπορεί να διαβιβάσει. Τα κράτη-μέλη, η Europol για παράδειγμα, απευθύνονται σε εμά για μια ανάλυση, για μια συγκεκριμένη περίπτωση και το κάνουμε. Γιατί ο βασικός στόχος είναι να μπορεί κανείς στη Eurojust να βρει ε, σε μία έρευνα ή σε μία ανάκριση τους κατάλληλους εταίρους, συνομιλητές. Ελπίζω να απάντησα κατά κάποιο τρόπο στην ερώτησή σας. Σε ό,τι αφορά τώρα την ερώτηση του κυρίου Βέμπερ για τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Eurojust, της κυρίας Βέμπερ μάλλον, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό απασχολεί πολλούς. Το βασικότερο πρόβλημα είναι η εξασφάλιση πληροφόρησης από τα κράτη-μέλη. Και ε, με τη νέα απόφαση για τη Eurojust νομίζω ότι έχει γίνει μεγάλη πρόοδος. Ε, βάσει το άρθρο 13 ε, υποχρεούνται τα κράτη-μέλη που έχουν ουσιαστικά διασυνοριακά ζητήματα σημαντικά να μας τα κοινοποιούν με συγκεκριμένου πολλού όρου και προποθέσει, αλλά αυτό είναι η κεντρική ιδέα. Να κοινοποιούν στη Eurojust ε, ε, εκρεμή ζητήματά του σε διασυνοριακό επίπεδο. Και εμεί μπορούμε να προσθέσουμε αξία εκεί με τι επαφέ που έχουμε και την οργάνωσή μα. Έτσι λοιπόν, ανταλλαγή ενημέρωση και πληροφόρηση παραμένει ζωτική σημασία για τη Eurojust. Επίσης αναφέρατε, κυρία Βέμπερ, ε, τα ε, κοινέ ανακριτικές ε, ερευνητικέ ομάδες και κατά πόσο προχωρούν γοργά στο έργο τους. Υπάρχουν και καλές ειδήσει. Δεν θέλω να με θεωρήσετε επιπόλαια αισιόδοξο, αλλά τα στοιχεία των κοινών ερευνητικών ομάδων βελτιώνονται. Μέχρι 1,5 χρόνο πριν Υπήρχε μεγάλη καχυποψία ε, των ενδιαφερομένων για τις κοινέ ερευνητικές ή ανακριτικές ομάδες. Το θεωρούσαν υπερβολικά γραφειοκρατικό, έτσι βαρύ ε, οικοδόμημα, εγχείρημα. Έχουν αρχίσει και αλλάζουν όμως οι νοοτροπίες. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι έχουν πλεονεκτήματα τέτοιες δομές και τις υιοθετεί. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ε, την επιτάχυνση που μπορούν να επιφέρουν αυτές οι ομάδες και την υπέρβαση ε, ορισμένων δυσκολιών που συνδέονται με διαφορετικά νομικά συστήματα και νομικούς πολιτισμούς. Αυτά. Ελπίζω να απάντησα σε ορισμένες από τις ανησυχίες σας. So um, ε, Σε ό,τι αφορά αυτά που είπε ο κύριος Γιακολίνο, πρέπει να σας πω ότι ο ρόλος της Eurojust, κοιτάξτε, είναι δεδομένος και πολύ συγκεκριμένη μια διάταξη που λέει όταν αυτό θεωρείται σκόπιμο μπορεί να ε, δώσει τη γνώμη της ε, Eurojust για την νομοθεσία ε, που αποφασίζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και όταν αυτό είναι σκόπιμο πραγματικά το κάνουμε και απευθύνονται σε εμάς, πηγαίνουμε στις Βρυξέλλες, στις συνεδριάσεις τους Τώρα για συγκεκριμένα για την εντολή ε, προστασίας που συζητούσατε προηγουμένως ή που αναφέρατε, μπορεί να μην είναι της αμέσου αρμοδιότητάς μας, αλλά προβλέπετε. Σε ό,τι ε, αφορά τώρα την ερώτηση που έκανε ο κύριος Μπρόνς ε, για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και κατά πόσο θεωρείται μια πράξη αξιόπινη σε μια χώρα και σε μια άλλη όχι. Είναι 32 κατηγορίες αδικημάτων αυτές. 32 κατηγορίες στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Είναι με απόφαση ε, πλαίσιο. Ε, η εκδίδουσα λοιπόν αρχή αν θεωρήσει ότι ε, μια αξιόπινη πράξη εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία τότε έχει εφαρμογή αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση ε, θα πρέπει να απαιτείται, να χαρακτηρίζεται αξιόπινη πράξη το αδίκημα και στις δύο χώρες. Ε, τώρα, για, όταν υπάρχουν, κύριε Δίας Δεμέρα, ε, διενέξεις για το ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο. Μα εκείνοι που είναι αρμόδιοι στα κράτη-μέλη, που έχουν το κύρος, ε, την εξουσία να αποφασίσουν, εκείνοι συμμετέχουν ε, στις συντονιστικές αυτές ε, επιτροπές και με παραδείγματα ας πούμε εάν ένας δικαστής στο βασίλειο της Ισπανίας ή ένας ε, δικαστής του Δικαστηρίου για την Τρομοκρατία της Αντίας National ενέχεται στην υπόθεση. Αυτό είναι ο συνομιλητής μα και μαζί θα αποφασίσουμε για το εάν και κατά πόσο θα πρέπει να ε, διωχθεί ε, σε ένα κράτος μέλος ε, ή σε ένα άλλο κράτος μέλος. Η περίπτωση αυτή. Αυτό λοιπόν εξαρτάται από τις εκάστοτε εξουσίες που έχει στο κράτος μέλος του ο κάθε δικαστής ή κάθε αρχή. Ελπίζω να απαντάει αυτό. Thank you. Ευχαριστώ πολύ κύριε Williams. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας και την ε, ε, προσπάθεια που καταβάλατε να συνοψίσετε. Έχουμε και την έκθεση ε, στα χέρια μας, κυκλοφόρησε. Ελπίζουμε να σας βλέπουμε συχνά σε τακτά χρονικά διαστήματα και προσβλέπουμε σε αυτό στην Επιτροπή Ελευθεριών. Ε, τέλειωσε ο χρόνος, αλλά έχουμε μια ανακοίνωση ακόμα. Ορισμός νέων εισηγητών. Μετά τη συνεδρίαση των συντονιστών, ορίστηκαν νέοι συντονιστές, ε, εισηγητές συγγνώμη, που είναι εξής. Ο κύριος Λούχαν για το Coin System. Η κυρία Φαγιόν, η συγγήτρια για την απελευθέρωση θεωρήσεων για τη Βοσνία και την Αλβανία και ο κ. Αλμπρέχτ, εισηγητής Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΠΑ για την προστασία των δεδομένων. Αυτοί είναι λοιπόν οι συγγητές Διακόπτουμε και επαναλαμβάνεται τη συνεδρίαση στις 3 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ.